Hello. Peter. Καλώς ήρθατε στην σημερινή συνεδρίαση. Η ημερήσια διάταξη είναι πολύ φορτημένη σήμερα. Οπότε θέλω να ξεκινήσουμε. Ίσως βέβαια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα αναγκαστώ να περιορίσω το χρόνο ομιλίας για να μπορέσουμε να εξετάσουμε όλα τα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Το πρώτο μας θέμα λοιπόν είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εγώ δεν έχω να προτείνω καμία τροποποίηση, αλλά όποιος έχει παρακαλώ, αν κάποιος έχει κάτι να πει. Όχι. Εγκρίνουμε λοιπόν την ημερήσια διάταξη. Καλώς. Ε, Τώρα, το επόμενο θέμα είναι τα πρακτικά, η έγκριση των πρακτικών δηλαδή, των συνεδριάσεων της 26ης Ιανουαρίου και της 10ης και 11ης Φεβρουαρίου. Εδώ λοιπόν, αν έχετε παρατηρήσεις ή σχόλια, εγκρίνονται τα πρακτικά, εγκρίνονται λοιπόν. Ωραία. Καλώ, συνεχίζουμε. Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Πρώτον. Βρίσκεται στο ίντερνετ η συνεδρίαση. Web streaming. Φαντάζομαι δεν έχετε πρόβλημα με αυτό. Ότι είμαστε στον αέρα. Τώρα για την αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη, 5 και 6 Φεβρουαρίου. Εγκρίνουμε την, ε, τα σχόλια που έχουμε εδώ, παρακαλώ. Yes, I just Πρόεδρε, ναι, αυτό που είπες ότι υπάρχει και εδώ πέρα μια αντιπροσωπεία ε, που σήμερα το πρωί μας έκαναν μια παρουσίαση στις Βρυξέλλες Έχουμε ένα σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη για τους εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών. Έχουμε λοιπόν μια τέτοια αντιπροσωπεία εδώ. Πρόεδρος, ναι, καλώς, καλώς ήρθατε. Εδώ, να παρακολουθήσετε τη συνεδρίασή μας. Να, η αντιπροσωπεία, εκεί πίσω. Καλώ. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Διαδικαστικό ακούσαμε από τον κύριο Κρήμα. Τώρα συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη και είμαστε στο σημείο 4. Δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Θα ψηφίσουμε σήμερα την έκθεση αυτή. Πριν όμω ξεκινήσουμε την ψηφοφορία θέλω βέβαια να δώσω το λόγο στον κύριο Μπρακέτο που είναι και ο εισηγητή. Δεν έχετε τίποτα να πείτε? Εντάξει, δεν σα αναγκάζουμε, όχι με το ζόρι. Ακούσατε τι είπα πριν για το χρόνο που μας πιέζει, οπότε σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πραγκέτο που δεν θέλετε το λόγο, οπότε θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Νομίζω ότι έχετε, ε, τις, ε, το, πήρατε μάλλον το μήνυμα για να έχετε τις κάρτες σας για την ψηφοφορία εδώ, έτσι δεν είναι. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτη τροπολογία είναι η τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και υπάρχει και ένα θέμα το οποίο ξέχασα να σας πω ότι συζήτησα το θέμα με τη γραμματεία για κάποιες τροπολογίες, κατά πόσο μπορούν να θεωρηθούν, να κρυθούν αποδεκτές ή όχι. Και διαπιστώσαμε ότι 24, 25, 26, 33 και 67, 67 όχι 66, αυτές οι τροπολογίες λοιπόν δεν μπορούν να κρυθούν αποδεκτές γιατί ανήκουν σε, ένα διαφορετικό, σε μια διαφορετική νομική βάση. Εντάξει, οπότε συνεχίζουμε τώρα. Συμβαστική α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Καταπίπτουν ε, οπότε κάποιες τροπολογίες με αποτέλεσμα να φτάνουμε στην τροπολογία 64. Υπέρ παρακαλώ της 64. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 τώρα. Υπέρ. 66 που είναι από τις αποδεκτές. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67 είπαμε δεν είναι αποδεκτή. 68 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να το ελέγξουμε αυτό με ηλεκτρονική ψηφοφορία. 71 λοιπόν. Ψηφίζουμε την 71 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 35 ψήφισαν. 17 υπέρ, 18 κατά. Συνεπώς, απορρίπτεται. 73 τώρα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω, αλλά επειδή δεν είναι τόσο σίγουρο το αποτέλεσμα, θα ελέγξουμε. Τροπολογία 73. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Όντω, δίκιο είχα. Ψήφισαν 38, 19 υπέρ, 19 κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. Αλλά όντω το αποτέλεσμα ήταν πολύ τσιματσιμό. Τώρα, τροπολογία 72 με προφορική τροπολογία για την ημερομηνία εφαρμογή του κανονισμού 883 κάθετος 2004. Με την προφορική αυτή τροποποίηση, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά και πάλι. Δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 39 ψήφισαν, 21 ψήφοι υπέρ, 17 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν. 74 με, με προφορική τροποποίηση. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12 και 75 έχουν αποσυρθεί, 76 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 80 υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 91 τώρα, τροπολογία 91. Εδώ έχουμε δύο τμήματα, κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα που ξεκινάει με το «Οι δημόσιες αρχές στα κράτη-μέλη» και τελειώνει με το υπό το άρθρο 18. Ψηφίσουμε λοιπόν αυτό το πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα τώρα. Το επόμενο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία Β υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτουν κάποιες τροπολογίες και φτάνουμε στη συμβαστική γάμα. Υπέρ παρακαλώ τη συμβαστική γάμα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. η 104 πίπτη. και έτσι ερχόμαστε στη συμβαστική δέλτα, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 105 έχει αποσυρθεί, 108 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 110. Με προφορική τροπολογία. Διαγράφονται οι γραμμές για τον ασθενή. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 111. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 113. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε καλύτερα. 114. Ελέγχουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 40 ψήφισαν, 19 ψήφοι υπέρ, 21 κατά. Καθόλου αποχές. Απορρίπτεται λοιπόν. Συνεχίζουμε. 116 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική ε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οπότε, περνάμε μετά από διάφορες τροπολογίες που καταπίπτουν στην 134 και 135 που είναι δύο τροπολογίες ταυτόσιμες. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 136 έχει αποσυρθεί. Κάποιες άλλες καταπίπτουν και έτσι φτάχνουμε στο σίγμα τάφ. Συμβαστική σίγμα τάφ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Καταπίπτουν με τα όλα μέχρι την 150. 150 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τώρα ζήτα G υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτουν δύο τροπολογίες και έτσι φτάνουμε στην 160. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 161. Με προφορική τροπολογία που έχει να κάνει με τον 883 κανονισμό 2004 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 163 έχει αποσυρθεί. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Συμβιβαστική H τα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν διάφορε 172 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 178 με προφορική τροπολογία που επίσης προσκαλούνται κλπ. Μέχρι τους συμμετέχοντες με προφορική τροπολογία. Λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 183 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 193 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 197 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα 198 εδώ έχουμε δύο τμήματα το πρώτο τμήμα που λέει ότι μετρήσει επιτρέπουν κτλ. Και, τελειώνει με την αυθεντικότητα της ηλεκτρονικής ε, συνταγολόγησης. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Λοιπόν, το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 201 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 202 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 203 υπέρ, κατά αποχές Εγκρίνεται. 204 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 205 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 26 τώρα. Αλλά αυτή δεν είναι παραδεκτή. 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ας την επαληθεύσουμε την ψηφοφορία αυτή λοιπόν ηλεκτρονικά την 30 Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρας. 40 ψηφίσατε, 21 υπέρ, 19 κατά και καμία αποχή εγκρίνεται επομένω. 4 υπέρ. Α, έχει αποσυρθεί αυτή. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 33 είναι μη παραδεκτή. Ποια ακολουθεί τώρα. Η 32 είχε απορριφθεί, ναι, ναι. Η 32 απερίφθη. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται υπάρχει μόνο 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τρία με μια προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα όπου αφαιρούνται οι λέξεις and entitlement to them, δηλαδή να έχουν αξίωση για το α ή β πράγμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 με μια προφορική τροπολογία υπέρ του ασθενούς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αυτή 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 24 και 25 είναι μη παραδεκτές. Φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία για το τροποποιημένο κείμενο και θα ψηφίσουμε εδώ ονομαστικά με τις ηλεκτρονικές κάρτες. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Το αποτέλεσμα είναι επί 41 ψηφισάντων, 35 υπέρ, 2 κατά και 4 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Μπαγκέτο. Για το κοινωνικό ταμείο τώρα. Okay. Då har vi kommit till eh, Ας προχωρήσουμε λοιπόν στο θέμα της επέκτασης των τύπων δαπανών που είναι επιλέξιμες και συνεισφορά από το ΕΚΤΑΦ. Μπορούμε να ψηφίσουμε, έχουμε δύο τροπολογίες. Την υπαριθμόν 1. Κύριε Στάουνερ, πριν να ψηφίσουμε και επειδή με έχει παρακαλέσει η κυρία Γκρέσλε επιθυμώ να πω ότι αποσύρει η κυρία Γκρέσλε τις δύο τροπολογίες της. Υπέροχα, λέει ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Άρα ε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Θα ψηφίσουμε την έκθεση την ίδια την έκθεση και το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου. Ας ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρας. Επί 40 ψηφισάντων 38 υπέρ 2 κατά και καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Κυρία Γιώργης. Ερχόμαστε στο επόμενο θέμα που είναι η κοινή πολιτική μετανάστευσης για την Ευρώπη, αρχές, ενέργειες και μέσα. Πρόκειται για γνωμοδότηση για την έκθεση της, Επιτροπή ε, Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Αρχίζουμε την ε, ψηφοφορία. Συμβαστική Α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 και 7 έχουν εκπέσει. 8 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι και εδώ χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε παρακαλώ. Πέρας. Επί 40 ψηφισάντων 18 υπέρ 22 κατά. Και καμία αποχή. Απορρίπτεται λοιπόν. Συμβαστική Β υπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και εδώ εκπίπτουν οι 9, οι 10, οι 11 δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Συμβαστική γάμα σε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προχωρούμε στην 15 υπέρ κατά 15 υπέρ κατά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 κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή και 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα ψηφίσουμε τώρα το σύνολο της γνωμοδοτήσεως όπως τροποποιήθηκε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ αρχίζει Ψηφίσατε παρακαλώ. Πέρας. Επί 39 ψηφισάντων, 37 υπέρ, μία ψήφος κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Μαντέιρα. Ερχόμαστε στο θέμα της κυρίας Παναγιωτοπούλου. για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των προσώπων που εκτελούν κινητές δραστηριότητες στις οδικές μεταφορές. Παρακαλώ. Uh, am dorit să vin uh, special la acest uh, vot. Sunt vicepreședinta din partea socialiștilor a Comisiei de Transport. Ήθελα να σας πω κύριε Πρόεδρε, λέει κυρία Τικάου. Α, μιλάει τώρα στα αγγλικά. Βρίσκομαι παρούσα εδώ ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, Μεταφορών και η στην ομάδα των Σοσιαλιστών. Η έκθεση αυτή είναι κρίσιμη σημασία για την ασφάλεια των οδικών μεταφορών και για την ασφάλεια των οδηγών. Πραγματικά έχει τεράστια σημασία και γι' αυτό παρακαλώ ιδιαίτερα όλους τους συναδέλφους να προσέξουν πώς ψηφίζουν. Είναι πάρα πολύ ε, σημαντική η έκθεση αυτή για όλους όσοι συμμετέχουν στις οδικές μεταφορές. Μάλλον δεν ήταν διαδικαστικό αυτό, κυρία μου, λέει ο πρόεδρος. Μπουζιλ Όντως δεν είναι διαδικαστικό και πιστεύω θα συμφωνήσετε και εσείς ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις. Ούτε αυτό ήταν διαδικαστικό βέβαια, απαντά ο πρόεδρος. Ε, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ. Θα προχωρήσουμε. περάσουμε στην ψηφοφορία. Πάμε στην τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 9. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 40 ψήφισαν, 23 υπέρ, 17 κατά. Καμία αποχή. Καταπίτη. Δεν συνεχίζεται η ψηφοφορία. Μια στιγμή. Uh, listen to me. Ακούστε όλοι σας θα πρέπει να ψηφίσουμε την νομοθετική πρόταση, που είναι κάτι το ίδιο. Θα ξεκινήσουμε ξανά, τα ίδια πάλι. Θα ψηφίσουμε λοιπόν την νομοθετική πρόταση. Δεν καταλαβαίνω γιατί λέει ο Πρόεδρος. Έχει απορριφθεί. I, Αν έχουμε διαφορετικές, διαφορετικές προτάσεις, τελικά τι περνάει ε, και διαφορετικά αποτελέσματα στην πληροφορία. Έχουμε ένα αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο αποτελέσματα και μάλιστα αντιφατικά μεταξύ τους. Was okay. nu nu European Τότε ας περάσουμε στο σημείο που αφορά το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την κατάρτιση. Όπως θα ξέρετε, υπάρχουν νέοι κανόνες για αυτό το, το ίδρυμα, για αυτόν τον οργανισμό. Έχουμε κάποιους καλεσμένους. Θα πρέπει να διορίσουμε κάποιους εμπειρογνώμονες για αυτό το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης. Έχουμε τρεις καλεσμένους που τους καλέσαμε μετά τη συνάντηση των συντονιστών. είναι εμπειρογνώμονες που πρότειναν οι συντονιστές. Αυτοί πρότειναν να διορίσει το Κοινοβούλιο. Τους καλέσαμε. Θα κάνουν κάποιες σύντομες δηλώσεις πριν περάσουμε στο διορισμό τους. Please, people here, all of you, some of you are very excited after. Ορισμένοι έχετε ταραχθεί από το αποτέλεσμα, το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα θα πρέπει να δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας. Παρακαλώ λοιπόν λίγη ησυχία. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Μεζιέ, Jean-François Μεζιέ, την κυρία Σάρα Πάρκιν, και τον κύριο Σταμάτη Παλοκρασά. Σας καλωσορίζω και τους τρεις. Κύριε Μεζιέ, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που με προσκαλέσατε σήμερα και πολύ σύντομα να αναφέρω δύο σημεία. Καταρχάς, ε, κατά την άποψή μου, ποιες είναι οι προτεραιότητες και η αποστολή του Ιδρύματος αυτού, όπως αναθεωρηθήθηκαν από τον κανονισμό του περασμένου Δεκεμβρίου και να σας εξηγήσω πώς εγώ προσωπικά αντιλαμβάνομαι μαζί με τους συναδέλφους τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουμε για να υλοποιήσουμε τις προσδοκίες της Επιτροπής σας. Η αποστολή και οι προτεραιότητες του Ιδρύματος καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην ε, ξανακάνουμε αυτά που έχουν ήδη γίνει και να αξιοποιήσουμε αντίθετα αυτά που έγιναν. Τρία σύντομα σημεία. Θα πρέπει να υπάρχει μια σφαιρική προσέγγιση της ε, διαβίου κατάρτισης, να προωθήσουμε δηλαδή το ανθρώπινο κεφάλαιο, τους ανθρώπινους πόρους και σε αυτή την ε, περίοδο κρίσης που διανύουμε είναι πολύ σημαντικό για να υπάρξει συνοχή κοινωνική και απασχολησιμότητα, να υπάρξει κατάρτιση των ατόμων. Και επίσης να έχουμε και τα κατάλληλα εργαλεία κατάρτισης ε, προς όφελος των εργοδοτών και των εργαζομένων. Επίσης θα πρέπει να μοιράζουμε μεταξύ μας τις πληροφορίες και τις αναλύσεις τα κράτη-μέλη, η Κομισιόν, αλλά και όλοι οι φορείς των ε, αποδεκτριών χωρών. Αυτό σημαίνει προετοιμασία για τις οικονομικές μεταλλαγές και μετασχηματισμούς και κυρίως μια συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι η σημασία ε, μιας αποτελεσματικής προσπάθειας όλων των εμπλεκομένων. Το Ίδρυμα δεν μπορεί να δουλέψει μόνο του, θα πρέπει να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των κρατών μελών, και των άλλων θεσμικών οργάνων όπως το ΣΕΝΤΕΦΟΠ ή του Ιδρύματος για το, του Δουβλίνου. Θα πρέπει να αναζητήσουμε αποτελεσματικές ε, συνεργασίες και να αποφύγουμε τη στήρα αντιπαράθεση και τον ανταγωνισμό. Δεύτερον, πώς θα εργαστούμε, πώς εγώ θεωρώ ότι θα υλοποιήσουμε την αποστολή που μας ε, εμπιστεύεστε. Πρώτο τμήμα, πρώτη πτυχή. Θα πρέπει να ακούμε αυτά που θέλει η Επιτροπή σας, να γνωρίσουμε πολύ σύντομα τις προτεραιότητές σας και τις ανησυχίες σας στον τομέα της κατάρτισης. Να δούμε τι διακυβεύεται από δημοσιονομικής απόψεως, να υπάρξει κοινωνικός διάλογος. Δεύτερο, δεύτερη πτυχή, να υπάρξει μια χρήσιμη συνεισφορά από μέρους μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος για την εφαρμογή των μεγάλων προγραμμάτων, της αξιολόγησής του, του προγράμματος και του προϋπολογισμού και στην ε, ανάλυση του απολογισμού και στην ε, αξιολόγηση της ε, εργασίας που έχει ήδη γίνει. Τρίτον, να είμαι σε επαφή με τους συναδέλφους, με την Επιτροπή σας και με τα διοικητικά όργανα του Ιδρύματος. Να σας ενημερώνουμε δηλαδή, να σας ρωτάμε, να σας κρούμε τον κόδωνα κινδύνου, ούτω ώστε να γνωρίζετε τι κάνει το Ίδρυμα, να υπάρχει δηλαδή λογοδοσία τακτική σωστή και μαζί με τους συναδέλφους, τους άλλους εμπειρογνώμονες, που να προωθήσουμε στο εσωτερικό του Ιδρύματος τα θέματα που σας ενδιαφέρουν, τα θεματικά, τα, τα γεωγραφικά. Θα ήθελα λοιπόν να βοηθήσω και εγώ να υπάρξει μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του Ιδρύματος και της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής σας για να είναι κανείς εμπειρογνώμονας θα πρέπει να κινητοποιεί και να χρησιμοποιεί όλη την εμπειρία που έχει. Θα διαβάσατε στο βιογραφικό μου τι εμπειρία έχω. Περιτώ λοιπόν να τα επαναλάβω όλα αυτά τα στοιχεία εδώ. Τα θέτω λοιπόν στην υπηρεσία σας και με αυτόν τον τρόπο ελπίζω να είμαι χρήσιμος και στην δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πάρκιν. Το λόγο έχει η κυρία Πάρκιν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ χαίρομαι που με προσκαλέσατε εδώ στην Επιτροπή σας σήμερα. Δεν θα επαναλάβω όσα μόλις ανέφερε ο συνάδελφος για το πώς θέλουμε να συνδεθούμε και να συνεργαστούμε μαζί σας. Νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο ότι καταρχάς θα πρέπει να φροντίσουμε να δούμε πώς θα πετύχουμε αυτά που θέλετε να πετύχουμε. Άρα θα πρέπει να συζητούμε μαζί σας. Ελπίζω να συνεργαζόμαστε σενά και να μπορέσουμε να, να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας και στις εξωτερικές σχέσεις για να υπάρχει πραγματικά καλή επικοινωνία. Να επικεντρωθώ σε αυτά που με απασχολούν ιδιαίτερα Έχω μεγάλη εμπειρία σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε κάποιους τομείς όπου στο Ηνωμένο Βασίλειο ενσωματώσαμε στοιχεία βιωσιμότητας. Συνεργαστήκαμε με επαγγελματικά σώματα και με επιτροπές από τον κλάδο για να δούμε πώς μπορούν να ενσωματέσουν νέους τομείς, νέες γνώσεις. Άρα, έχω κάποια εμπειρία στο τομέα αυτό. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω ότι υπάρχει αυτή η επέκταση της ιδέας της επένδυσης στον ανθρώπινο κεφάλαιο και της ευρύτερης εντολής του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την επαγγελματική κατάρταση. Όπως είπε και ο συνάδελφος, ε, ο επόμενος καιρός θα είναι πάρα πολύ δύσκολος και νομίζω ότι αν κάνουμε αυτή τη σύνδεση μεταξύ των ικανοτήτων, των γνώσεων και της δυνατότητας εξέβρεσης εργασίας, αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια πολιτικά δύσκολη κατάσταση. Άρα εγώ θα μπορέσω να συμβάλλω λόγω της εμπειρίας μου με τη συνεργασία με κυβερνητικά σώματα αλλά και με τον ίδιο τον κλάδο, όπως για παράδειγμα τον κλάδο του τουρισμού, προκειμένου να πετύχουμε αυτό που πιστεύω ότι επιδιώκεται μέσω της σχέσης αυτής. Κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω τώρα. Τα γαλλικά μου είναι καλά, αλλά έχω και εμπειρία σε ό,τι αφορά τις αναδυόμενες δημοκρατίες, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στο συγκεκριμένη ιδιότητα προκειμένου να εφαρμοστούν τα προγράμματα που θέλει να εφαρμόσει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης και σε ό,τι αφορά την ενημέρωσή σας για ενδεχόμενα προβλήματα. Και έχω πολλή εμπειρία σε ό,τι αφορά την ε, διακυβέρνηση, διαχείριση πολιτικών σωμάτων. Και μπορώ να συμβάλλω λοιπόν με την εμπειρία μου αυτή. Σας ευχαριστώ. Och ευχαριστώ. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ μαζί με τους δύο συναδέλφους. Πέρα από τις ερωτήσεις που μας ε, θέσατε σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος ε, για την κατάρτιση και του Διοικητικού του Συμβουλίου να σας πω ότι το Ίδρυμα στο πλαίσιο της αποστολής του, αν δεν το έχει ήδη κάνει, θα πρέπει να αναθεωρήσει τις προτεραιότητες του και την συνολική του στρατηγική σε ό,τι αφορά την παγκόσμια ύφεση και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και σε ό,τι αφορά τα συστήματα απασχόλησης και απασχόλησης. Αυτό θα πρέπει να γίνει από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την κοινωνική ατζέντα εν ώψη της κρίσης. Για παράδειγμα, το σύστημα, μάλλον το σύστημα κατάρτισης εξακολουθεί να αποτελεί το σωστό μέσο για την καταπολέμηση της ανεργίας και της ύφεσης στα κράτη-μέλη. Ίσως χρειάζεται ένα άλλο είδος κατάρτισης, ιδιαίτερα υπό τις ακραίες ε, συνθήκες μαζικών απολύσεων και μαζικής ανεργίας, σε ό,τι αφορά τον ρόλο που θα αναλάμβανα εγώ ως εμπειρογνώμονας διορισμένος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικεντρώνεται κυρίως στις κοινωνικές πτυχές της απασχόλησης και της κατάρτισης. Και άρα ο εμπειρογνώμονας, οι εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Ίδρυμα θα πρέπει να τονίζουν τα κρίσιμα αυτά ζητήματα που αφορούν τις κοινωνικές πτυχές της απασχόλησης και κατάρτισης, όπως για παράδειγμα οι ίσες ευκαιρίες, ευκαιρίες ε, ε, εκ νέου κατάρτισης, εγκατάλειψης του σχολείου, διευκόλυνσης ε, των όσων αναζητούν εργασία και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν με την Επιτροπή πέρα από τις σημαντικές οδούς επικοινωνίας. Θα μπορούσα να καλύπτω τις ανάγκες ενημέρωσης ε, της ε, Επιτροπής σας αναφορικά με τις δραστηριότητε του Ιδρύματος και σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων οι εμπειρογνώμονες και ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής θα μπορούσαν να συζητούν ιδιαίτερα έγγραφα, για παράδειγμα έγγραφα πολιτικής και συγκεκριμένες ανάγκες. Για να συζητούνται κρίσιμα θέματα για το Ίδρυμα και για την Επιτροπή προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία αναθεώρησης της εντολής του Ιδρύματος. Σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ μάλλον. Ακούσαμε τους τρεις ομιλητές πριν από κάποιο διάστημα, πριν από ορισμένες συνεδριάσεις είχαμε παρουσία εδώ των διαφόρων οργανισμών και του Ιδρύματος. Έχουμε καλή συνεργασία με το Ιδρύμα αλλά και με άλλους οργανισμούς και ελπίζουμε να συνεχιστεί η καλή συνεργασία και με εσάς το θέμα της εκπαίδευσης θα λαμβάνει όλο και μεγαλύτερη σημασία στην κοινωνία εν ώψη των οικονομικών εξελίξεων που καθιστούν απαραίτητο και τον καθένα να βελτιώνει την κατάρτισή του διαρκώς, ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσεων όπως είπε κάποιος από εσά και σίγουρα υπάρχει η δυνατότητα και μέσα σε περίοδους κρίσεων να βελτιώνονται κάποιες ικανότητες, κάποια προσόντα που ίσως δεν γίνεται πάντοτε σε περίοδους ευίωνης οικονομικής συγκυρίας. Θα απευθύνω τώρα τον, το ερώτημα στην Επιτροπή. Έχουμε τρεις εμπειρογνώμονες, έχουμε συζητήσει και μεταξύ των συντονιστών, τον κύριο Μεζιέρ, την κυρία Πάρκιν και τον κύριο Παλαιοφρασά. Συμφωνείτε όλοι ότι τα τρία αυτά πρόσωπα θα είναι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου. Δεν φαίνεται να, έχει, να υπάρχει κανένας, καμία ένσταση. Είστε λοιπόν, εκλέγεστε λοιπόν εκπρόσωποι στην, του Κοινοβουλίου στην, ε, στο Ίδρυμα. Μπορείτε να παραμείνετε στην αίθουσα αν επιθυμείτε θα συνεχίσουμε με το θέμα του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης. Δεν είσαι όμως υποχρεωμένοι να παραμείνετε. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα που είναι η τροποποίηση του κανονισμού 1927-06 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Θα δώσω πρώτον λόγο στην κυρία Στάουνερ. Ωστόσο, ο συνονόματός μου Γιάνν Όλσον δηλαδή που μαζί μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα φύγουμε κιόλα, θα λάβει και αυτό το λόγο. Πάντω πρώτα η κυρία Στάουνερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για την τροποποίηση του κανονισμού του ε, Ταμείου Παγκοσμιοποίησεως, το οποίο, θέμα το οποίο συζητήσαμε. Οι, κατέστησαν σαφείς οι διάφορες διστάμενες απόψεις, έχουν υποβληθεί και σχετικές τροπολογίες που κυρίως αναφέρονται στα πλέον επίμαχα θέματα έναν πιο συγκεκριμένο ορισμό ε, των αιτιών χρηματοδοτήσεως, δηλαδή τον ορισμό, ε, τέλος πάντων τι είναι παγκοσμιοποίηση με απλά λόγια το ε, χρονικό διάστημα που πρέπει να γίνεται η απαλλαγή επίσης τις διάφορες παροχές τις διάφορες προθεσμίες, το κόστος, ε, το συνοδευτικό κόστος κλπ. Η Κομισιόν προτείνει 35, εγώ προτείνω 25, υπάρχουν και άλλες προτάσεις για πιο χαμηλά ακόμα. Η χρηματοδότηση, το ύψος χρηματοδότησης από πλευράς Κομισιόν, η οποία έχει προτείνει 75% επίσης εκεί ε, δίστατη απόψεις γιατί υπάρχουν άλλες προτάσεις για υψηλότερες, ε, υψηλότερα ποσοστά και βέβαια και το χρονικό διάστημα εκτέλεσης. Η Επιτροπή θέλει 24 μήνο και εγώ νομίζω ότι εν ώψη του ότι οι παροχές αυτές δεν μπορεί να είναι διαρκείς θα πρέπει και το διάστημα να είναι συντομότερο σημαντικά συντομότερο. Αυτά είναι τα βασικότερα σημεία στα οποία αναφέρονται οι τροπολογίες. Η δική μου διαδικαστική πρόταση θα ήταν τώρα να κάνω μια προσπάθεια προσέγγισης σε ορισμένα θέματα. Θα έρθω σε επαφή και με τις άλλες πολιτικές ομάδες και με τους τροπολογούντες. Ε, όμως πιστεύω ότι σε ορισμένα δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε, δεν πρόκειται να τα βρούμε. Έτσι έχουν τα πράγματα για την ώρα. Ίσως οι ε, συνάδελφοί μου που έχουν κυρίως καταθέσει τροπολογίες να λάβουν το λόγο να εξηγήσουν με περισσότερη λεπτομέρεια το τι επιθυμούν. Σωστά, λάθος κουμπί Ε, πριν δώσω τον λόγο στα μέλη της Επιτροπής, Θέλω να δώσω πρώτα τον λόγο στον κύριο Γιάνν Όλσεν της ΕΚΟΣΟΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνει το δικαίωμα να ομιλήσω εξ ονόματος ε, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Έχω στα αγγλικά κάνει τις σημειώσεις μου και αυτό θα συνεχίσω στα αγγλικά. Από τη, δική, από μας πλευρά έχουμε υποβάλει σχέδιο γνωμοδοτήσεως το οποίο σας έχουμε διαβιβάσει. Δύο μικρές αλλαγές για την τροποποίηση που, που προτείνεται για τον Ιούνιο του 2010 και που έχει ως στόχο να γίνει ένα είδος απογραφής του Ταμείου. Αυτό όμως δεν θα είναι δυνατόν. Άρα δεν θα κάνουμε αυτή την επιλογή. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να γίνει μια αναθεώρηση για, μέσα στον επόμενο ένα ή ενάμιση χρόνο. Έχουν προτείνει επίσης να προβλεφθεί ένα δις ευρώ αντί για τα 500 εκατομμύρια που προβλέπονται για την ώρα. Ένα δισεκατομμύριο λοιπόν. Για την ώρα δεν φαίνεται να ε, μπορεί αυτό να γίνει αντικείμενο συμφωνίας. Ωστόσο, η πρόταση κανονισμού λέει ότι το, οικονομικό, το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Σχέδιο Ανοικοδόμησης θα προβλέπει και εφαρμογή των υποναθεώρηση κανόνων. Εμείς πάντως είμαστε υπέρ της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογή του Ταμείου της Παγκοσμιοποίησης λόγω και της σοβούς οικονομικής κρίσης. Ε, θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να μειωθεί το νούμερο από χίλιους σε πεντακόσους απολυόμενους ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει το Ταμείο. Θεωρούμε επίσης ότι στο άθρο 8Γ προβλέπεται στον κανονισμό, μας, στον κανονισμό του Ταμείου μάλλον ε, προβλέπεται ότι από ορισμένε περιστάσεις όπως μικρές αγοράς, αγορές εργασίας το μέγεθος αγοράς εργασίας μπορεί να αποτελέσει επιχείρημα για την χρήση των πόρων του Ταμείου και για λιγότερες από 500 απολύσεις. Σίγουρα είμαστε ε, σύμφωνοι να κατέβει κάτω από τους 24 μήνες η ε, συμμετοχή της κοινότητας να είναι της τάξης του 75% και ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει οι κοινωνικοί εταίροι να παίξουν ενεργό ρόλο στην διαχείριση του Ταμείου, να ζητείτε η γνώμη τους και, στις, ε, και στην περίοδο της διαδικασίας για την υποβολή αιτήσεως. Και γι' αυτό έχουμε προτείνει και εμείς τροπολογίες στο άρθρο 5.2 και προτείνουμε και προσθήκη νέας παραγράφου που να λέει ότι επειδή είναι ουσιώδου σημασία η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, οι ε, αιτήσει που θα υποβάλλονται ε, να γίνονται αντικείμενο διαβούλευση και με του κοινωνικού εταίρους. Και για την τεχνική αρρωγή ε, θεωρούμε επίσης ότι είναι σημαντική. Προτείνουμε λοιπόν νέα παράγραφο 4 που να λέει περίπου τα εξή ότι η τεχνική αρρωγή θα πρέπει να έχει ενεργό χαρακτήρα και να ε, εμπλέκονται και οι χώρες μέλη και οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι. Προσωπικά λοιπόν και μάλιστα και αν δεν, ακόμα και αν δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση εγώ θα πρότεινα να αυξηθεί στο 0,4 η ε, τεχνική αρρωγή. Τελευταία παρατήρηση θεωρούμε ότι το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα στα διαρθωτικά ταμεία ώστε και οι περιφερειακές αρχές και οι κοινωνικοί εταίροι και οι διάφορες ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κτλ. να συμβάλλουν και αυτοί με τον τρόπο τους στην εφαρμογή του ε, Ταμείου Παγκοσμιοποίησης και ε, τον συντονισμό του με τις δράσεις κυρίως του Κοινωνικού Ταμείου. Σας ευχαριστώ. Ταξιμιουκέ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχω εδώ τον κύριο Λίντε, Κοντινή, ρέτερ και Λίντ. Ο κύριο Λίντε πρώτα. Παρακαλώ κύριε Λίντε. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πρόεδρε, η ομάδα μου έχει ορίσει δύο σκιώδεις εισηγητές έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τουλάχιστον ένας από τους δύο θα ήταν παρόν. Αλλά να, που κανένας από τους δύο δεν είναι παρόν. Εκ μέρους τους πάντως θα μιλήσω. Ε, οι συνάδελφοι Ντιπουή και είναι εδώ πέρα στη διάθεσή σας για συζήτηση στη συνέχεια. Λοιπόν, δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα η ομάδα μου επιθυμεί να στηρίξει την πρόταση της Επιτροπής. Μας φαίνεται ότι αντιστοιχεί στις ανάγκες που υπάρχουν. Έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, υποστηρίζοντας αυτή την αρχική πρόταση, έχουμε την τάση να απορρίψουμε τροπολογίες. Είτε αποδυναμώνουν την πρόταση αυτή, είτε την αλλάζουν. Εμείς θέλουμε να μείνει ως έχει η πρόταση της Επιτροπής, να μην αλλάξει. Εννοείται ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και με τον εισηγητή και με τις άλλες πολιτικές ομάδες, αλλά σας λέω ότι καταρχήν αυτή είναι η στάση της ομάδας μου. Απριόρι σκοπεύουμε να κρατήσουμε αυτή τη γραμμή και στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, παρακαλώ. Κοτεινή Σρότερ. Κοτεινή. Κοτεινή πρώτα. Πρόεδρε, ευχαριστώ λέει ο κύριος Στην ε, προηγούμενη συνεδρίαση που είχαμε, εγώ είχα πάρει το λόγο για πολύ. Σήμερα θα φροντίσω να μην μιλήσω τόσο πολύ. Αλλά είχαμε βγει από τη συνεδρίαση αυτή λέγοντας ότι χρειαζόμασταν ψήφισμα. Και τώρα μόλις μας έγραψε ο κύριος το ψήφισμα. Ακριβώς. Αυτό είναι για την αναθεώρηση που θέλουμε μετά από ένα χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ και εγώ με τον προλαλήσαντα ότι δηλαδή και εμείς θέλουμε να παραμείνουμε στην στη θέση της Επιτροπής και να μην την αλλάξουμε. Αν χρειάζεται τώρα ε, αλλαγή, ανακαίνιση, ναι ασφαλώς χρειάζεται αλλαγή. Έπειτα η συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση είναι σημαντική γιατί πρέπει να ανταποκριθούμε με κάποιο τρόπο στην κρίση. Έπειτα, αν θέλουμε εξυγχρονισμό του Ταμείου. Ναι, και μάλιστα είπατε ότι οι δικές μας προτάσεις είχαν χρησιμοποιηθεί την προηγούμενη φορά. Τέταρτον, άλλες αλλαγές θα μπορούσαν να προβλεφθούν. Ναι, λέω και εδώ, γιατί στην έκθεση και στις τροπολογίες που έχουν κατατοθεί φαίνεται αυτό. Και είχαμε πει ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για ψήφισμα και να το ψήφισμα μας το έγραψε ο κύριος με αυτά που είπε. Έπειτα, είναι επιθυμητό να τροποποιήσουμε την πρόταση της Επιτροπής και εδώ συμφωνώ μαζί σου. Όχι. Διότι επιβραδύνεται τότε η διαδικασία και κινδυνεύουμε να χάσουμε τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Γι' αυτό λοιπόν εγώ και προτείνω στην ομάδα μου να ακολουθήσουμε την Επιτροπή, να μείνουμε στην πρόταση του κυρίου που κάνει ένα πολύ καλό ψήφισμα και έπειτα ε, το ταμείο το χρειάζονται οι εργαζόμενοι και γι' αυτό πρέπει σε πρώτη ανάγνωση να περάσει. Ευχαριστούμε, Σα Σας ευχαριστώ. Εγώ πιστεύω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Επειδή δεν είναι σαφές κατά πόσο τα κονδύλια αυτά τα επιπρόσθετα θα χρησιμοποιηθούν με βιώσιμο τρόπο. Δηλαδή, αν υπάρχουν σωστά κριτήρια. Εμείς θέλουμε βιώσιμη χρήση των κονδυλίων αυτών. Θέλουμε να υπάρχει μετακπαίδευση για όσους έχουν απολυθεί, όχι απλά να απολύονται και να παίρνουμε τα λίγα χρήματα και εκείνη τελειώνει η ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν ε, προσδώσαμε μία, έναν προσανατολισμό για το ποια κατεύθυνση θα πρέπει να λάβουν τα κονδύλια αυτά και δηλώνουμε ότι καλό θα ήταν να προσθέσουμε αυτή την κατεύθυνση αυτή στο κείμενο για να καταστεί σαφές ότι υπάρχει κάποιος απότερος στόχος στην, ε, στα κονδύλια αυτά. Όχι δηλαδή απλά να πάρουν για κάποιο χρονικό διάστημα κάποια χρήματα και μετά τίποτα. Να υπάρχει μία σωστή μετακπαίδευση. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά νέους επαγγελματικούς προσανατολισμούς. Νομίζω ότι η, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι προβληματική σε ό,τι αφορά την τεχνική αρρωγή, γιατί δεν είναι σαφές ότι αυτό χρειάζεται, γιατί όλα τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας μας καταδεικνύουν ότι όπου θεωρούσαμε ότι υπήρχε υπερβολική τεχνική βοήθεια, τελικά ήμασταν κάτω από το όριο του κανονισμού. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής είναι απαράδεκτη. Και εδώ θα υποβάλουμε βέτο πραγματικά, γιατί αυτό η επιπρόσθετη τεχνική, τεχνητή, τεχνική αρρωγή ουσιαστικά υποφελεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν είναι αυτό ο στόχο. Ο στόχο είναι να ωφελήσει του εργαζόμενου. Ένα άλλο πρόβλημα είναι τι σχέση υπάρχει με το ESF σημαντικός και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Γι' αυτό θέλουμε το ποσοστό χρηματοδότηση να είναι ακριβώς το ίδιο όπως και στο ESF. Γιατί δάλλως θα υπάρχουν μεγάλες ενοχλήσεις, μεγάλες ε, διαστρεβλώσεις, αν υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες σε ό,τι αφορά την τεχνική προσαρμογή. Δεν συμφωνούμε λοιπόν με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και όπου χρησιμοποιούνται τα ESF ε, υπάρχουν προβλήματα. Εμείς θέλουμε να ωφεληθούν οι εργαζόμενοι. Η εισηγήτρια δεν έχει λάβει ακόμα θέση για τις τροπολογίες μας και αυτό εμάς μας ανησυχεί. Αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί και να αποδεχτεί τις προτάσεις μας. Γιατί για μας αυτό θα είναι καθοριστικό για το κατά πόσο θα υποστηρίξουμε ή όχι την έκθεση. Πολύ. Uh, yes, thank you. Η κυρία Λίν, ευχαριστώ. Και εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις για το χρονοδιάγραμμα. Γιατί αλλάζοντα ε, το ταμείο, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών. Έχουμε δει τέτοιες απώλειες θέσεων απασχόλησης που βλέπουμε ότι χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω. Νόμιζα ότι είχαμε συμφωνήσει ότι δεν θα κατατεθούν τροπολογίες για να περάσει. Εφόσον όμως έχουν κατατεθεί τώρα τροπολογίες, μήπως κάποιος θα μπορούσε να μας δώσει κάποια ιδέα πώς θα προχωρήσουμε με το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή σε πρώτη ανάγνωση δεν έχουμε συμφωνία, τι θα γίνει διότι με τις καταστροφές που αντιμετωπίζουμε όλες τις χώρες μας, εξαιτία της οικονομικής κρίσης, είναι πολύ σημαντικό να περάσει αυτό το ταμείο σε γίνεται πιο γρήγορα. Συνήθω δεν μου αρέσει να έχουμε συμφωνίε στην πρώτη ανάγνωση. Πιστεύω ότι η συνδιαλλαγή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να ακουστεί η φωνή του Κοινοβουλίου. Αλλά εδώ, για αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση που τα χρειαζόμαστε τα χρήματα, πρέπει να ξέρουμε με τι ρυθμού θα προχωρήσουμε μετά. Θα μπορούσε κάποιο να μα καθοδηγήσει λίγο να μας πει πώς θα πάνε τα πράγματα μετά. Πρόεδρος, πριν δώσω το λόγο στην Επιτροπή, αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής, ότι θα ψηφίσουμε 31 Μαρτίου και μετά θα ξέρουμε τη θέση της Επιτροπής μας και θα δούμε κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε σε πρώτη ανάγνωση. Αν όχι, ε, δεν θα έρθουν τα χρήματα τόσο γρήγορα. Ναι, όχι αυτή τη Δευτέρα, ναι. Την επόμενη. Πάντως, στην επόμενη συνεδρία θα ξέρουμε. Έτσι καλώς ακούτε τη συζήτηση, μπορείτε να βγάλετε κάποια συμπεράσματα για το ποια είναι η πλειοψηφία. Έτσι, παρακαλώ κύριε Στάνο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση γιατί η γνωμοδότηση μου είναι πολύ... Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή. Θα ήθελα όμως να μας διευκρινίσετε κάποια πράγματα. Πώς τοποθετείτε σε μία τόσο πολύπλοκη κατάσταση αναφορικά με την επιδότηση και πώς φαντάζεται ότι θα συμμετέχουν και οι κοινωνικοί εταίροι. Το δεύτερο νομίζω το έθιξε ήδη και η κυρία Σρέντερ. Αν θέλουμε το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης να συμπληρώσει το Ταμείο το κοινωνικό, εγώ έχω προβλήματα, έχω κάποια προβλήματα και έχω κάνει και κάποιες τροπολογίες αναφορικά με αυτά. Θα πρέπει να αντιληφθούμε αγαπητοί συνάδελφοι ότι όλα όσα ξοδεύουμε στο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης ουσιαστικά αφαιρούνται από το Ταμείο το κοινωνικό. Και είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι το πολύ καλό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι το Ταμείο το κοινωνικό. Αυτό λειτουργεί πραγματικά πολύ σωστά αποτέλεσε και το πρώτο εργαλείο που είχαμε στη διάθεσή μας και πραγματικά πετυχαίνει τις πολιτικούς μας στόχους. Δεν έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι συμβαίνει το ίδιο και με στο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή, ουσιαστικά από ένα πολύ καλά συντονισμένο εργαλείο παίρνουμε και αφαιρούμε τα κονδύλια. Θεωρώ ότι το κοινωνικό ταμείο θα έπρεπε να παραμείνει το βασικό εργαλείο, γιατί είναι και βιώσιμο και επιτυγχάνει τους στόχους του και το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να είναι ένα προσωρινό εργαλείο, το οποίο σε καμία περίπτωση θα πρέπει να παραμερίσει το κοινωνικό ταμείο. Γι' αυτό λοιπόν ε, μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι με τόσο χαλαρά κριτήρια υπονομεύεται το κοινωνικό ταμείο. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Αυτά ήταν τα δύο στοιχεία που ήθελα να θίξω και το ανέφερα επειδή το είπε και η κυρία Σρόιντερ. Έχω την εντύπωση ότι με τις τροπολογίες της συναδέλφου Σρόιντερ μπορώ να θεωρήσω ότι ικανοποιούμαστε κι εμείς. Ικανοποιείται η θέση μας. Και εγώ είμαι κατά της αύξησης της τεχνικής αρρωγής. Γιατί όπως είπε και η συνάδελφος Φρόντερ, τα κονδύλια αυτά εφελούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά από πέντε χρόνια στην Επιτροπή Προπολογισμών δεν χρειάζεται να σας αναλύσω τι προβλήματα αντιμετωπίσαμε ε, με την τεχνική αρρωγή τα έτη 99 2004, εγώ θέλω τα χρήματα αυτά να ωφελήσουν αυτούς για τους οποίους προορίζονται, όχι τους υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και επίσης ε, θεωρώ ότι προβληματικό είναι και το θέμα της αύξησης της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το 75% ή ακόμα και παραπάνω της 100% όλα αυτά που αναφέρονται αλλά μου αρέσουν και οι τροπολογίες που αναφέρονται στην διευκρίνηση των ε, επιδόσεων. Νομίζω ότι οι εμπειρίες των τελευταίων ετών μας οδηγούν σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα και συμπέρασμα. Δεν μπορούμε να παραμένουμε στις ε, κλασικές, στα κλασικά ε, στις κλασικές επιδοτήσεις, στα κλασικά επιδόματα. Θα πρέπει να τα ορίσουμε όλα αυτά με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Στάουνερ, νομίζω ότι θα έπρεπε να συνοψίσετε τη συζήτηση. Αλλά τελικά εσείς θέσατε ένα ερώτημα με την παρέμβασή σας. Δεν ξέρω αν ο κύριος Όλσεν θέλει το λόγο. Ναι, ο κύριος Όλσεν και συνεχεία και η Κομισιόν μου κάνει νόημα ότι θέλει το λόγο. Ίσως να υπάρχει μια παρανόηση, κυρία Στάουνερ. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι το Ταμείο παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα πρέπει να είναι ένα συμπλήρωμα. Δεν θα πρέπει να κάνει ξανά τη δουλειά που κάνει το Κοινωνικό Ταμείο. Θα πρέπει να είναι κάτι το παραπάνω. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο παίζει το ρόλο του και οι κοινωνικοί εταίροι μπλέκονται στην όλη διαδικασία. Για το θέμα των κοινωνικών εταίρων μάλιστα, οι κοινωνικοί εταίροι είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να συμμετάσχουν στην ε, διαχείριση της όλης προσπάθειας. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η τεχνική αρρωγή είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εμπλέκονται οι κοινωνικοί εταίροι στην όλη προσπάθεια. Κύριο Γιώργενσεν, θα πρέπει να κάνω δύο διευθυνιστικές παρατηρήσει. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την προέλευση των χρημάτων του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης, αναφέρθηκε ότι παίρνουμε χρήματα από το Κοινωνικό Ταμείο και τα χρησιμοποιούμε για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Αυτό είναι λάθος. Με βάση τη διαθεσμική συμφωνία που διέπει το Ταμείο ε, Παγκοσμιοποίησης και τον προϋπολογισμό του μπορούμε να πάρουμε χρήματα ε, που δεν θα δαπανώνε οπουδήποτε στο προϋπολογισμό, σε οποιαδήποτε γραμμή του προϋπολογισμού, εκτός από τα χρήματα του Κοινωνικού Ταμείου. Επομένω είναι λάθος και παραπληροφόρηση το γεγονός ότι παίρνουμε χρήματα από το Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο, την τεχνική αρρωγή που προτείναμε. Μια παρατήρηση για αυτή. Πιστεύουμε ότι ξεκαθαρίσαμε ποιο είναι το πλαίσιο της πρότασης αυτής. Χρειαζόμαστε κάποια χρήματα, όχι πολλά, αλλά κάποια χρήματα, ούτω ώστε να υπάρχει μια γνώση για τις μαζικές απολύσεις. Πρόκειται για γνώσεις εντελώς διασκορπισμένες, ε, εντελώς διάσπαρτες. Ε, θα πρέπει να έχουμε πολύ πιο συνεκτικές ε, πληροφορίες για τις μαζικές απολύσεις στην πρόταση έχουμε βάλει ότι η Κομισιόν δεν κάνει ό,τι θέλει. Θα σας προτείνουμε σε εσά και στο Συμβούλιο οτιδήποτε πριν από κάθε δημοσιονομικό έτος τι μπαίνει στην τεχνική αρρωγή, τι κονδύλια πάνε για την τεχνική αρρωγή και εσείς αποφασίζετε λοιπόν εάν το έτοιμά μας είναι σωστό και συνάδει με τον κανονισμό. Επομένως νομίζω το έχουμε καλύψει και αυτό το θέμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρος, ωραία, ευχαριστώ. Νομίζω ότι κλείνει η συζήτηση εδώ για το σημείο αυτό. όπω είπα και προηγουμένω, θα ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση για το σημείο αυτό στι 31 δηλαδή Μαρτίου. Επομένως θα ξέρουμε μέχρι τις 31 Μαρτίου τι γνώμη έχει η Επιτροπή και θα, είμαστε, θα έχουμε ξεκαθαρίσει τα πράγματα για το αν θα μπορούσαμε δηλαδή να φτάσουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Τελείωσε η συζήτηση για αυτό το σημείο και πάμε στο σημείο 10 της σημερινής διάταξης τώρα. Ε, μέτρα για να βελτιώσουμε την ασφάλεια ε, στο χώρο εργασίας για τις έγκυες ε, γυναίκες, για τις λεχόνες και τις θυλάζουσες ε, μητέρες. Η κυρία Μαδέρα έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν σας πω οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί είναι κρίμα που δεν έχουμε την πρωτότυπη εκδοχή των τροπολογιών, το original δηλαδή των τροπολογιών για να δουλέψουμε πιο σωστά. Δουλεύουμε πάνω σε μεταφράσεις που δεν είναι επίσημες, όλες τουλάχιστον. Μπορούμε να δουλέψουμε, αλλά δεν είναι ο καταλληλότερος τρόπος. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν για αυτόν τον λόγο. Και δεν νομίζω ότι είναι και σωστό για όλους τους συναδέλφους, ακόμη και για μένα, που είμαι εισηγήτρια, για τη δική μου γλώσσα δηλαδή. Δεν δουλεύουμε επίσημη μετάφραση. Τέλος πάντων, τούτου λεχθέντος, η δουλειά μας διευκολύνεται από το γεγονός ότι συμφωνούμε για τις περισσότερες τροπολογίες. Δεν συνάντησα μείζωνα προβλήματα για τις τροπολογίες. Το θέμα που μας απασχολεί σήμερα είναι το θέμα των δικαιωμάτων, της προστασίας στον χώρο εργασίας. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος κοινός παρανομαστής ε, στην Ευρώπη. Θα πρέπει να συμφωνούμε με τις προδιαγραφές του του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εργασίας και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται εδώ. Νομίζω ότι όλες οι τροπολογίες οι οποίες παρουσιάστηκαν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Έχω όμως για κάποιες, ε, κάποιες αμφιβολίες. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία Shredder, θα μπορούσε η κυρία Σρέντερ να μας εξηγήσει τις τροπολογίες 21 και 58. Έχω κάποιες αμφιβολίες σε ό,τι αφορά την ε, ερμηνεία των στόχων. Για τις τροπολογίες 35 και 38 της κυρίας Βάισπέργκερ, ίσως δεν τις κατάλαβα καλά. Δεν κατάλαβα καλά τις προθέσεις της κυρίας Βάισμπεργκερ. Αλλά η κυρία Βάισμπεργκερ δεν είναι παρούσα και δεν μπορεί να με βοηθήσει. Όμως ίσως η κυρία Σρέντερ θα μπορούσε να μας δώσει μια εξήγηση για τις τροπολογίες 21 ε, και 58. Τι επιδιώκεται με αυτές τις τροπολογίες ακριβώς, κυρία Σρέντερ. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε αν η ε, κυρία Σρέντερ μου δώσε τις απαραίτητες εξηγήσεις. Αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντα πολύ εύκολο να παρουσιαστούν ε, συμβιβαστικές ε, τροπολογίες. Αλλά η προσέγγιση μεταξύ μας, για την οποία έκανα λόγο προηγουμένως, ε, είναι ένα θέμα αρκετά λεπτό και αφορά όλες τις πολιτικές ομάδες. Μέσα σε ένα χώρο ευρωπαϊκό μεγάλης κινητικότητας ό,τι αφορά την εργασία, είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ένα ελάχιστο βαθμό δικαιωμάτων, κάποια ελάχιστα δικαιώματα και να συμμορφωνόμαστε με τα όσα απαιτεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εργασίας. Αν θα μπορούσε η Προεδρία να μας βοηθήσει λίγο εδώ, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε πολύ πιο γρήγορα Κοινοβούλιο και Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Τρία άτομα, κυρία Λίν, κυρία Σόντερ και κυρία Στάουνερ. Κυρία Λίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποθέτω ότι τότε δεχόσαστε την δικιά μου, την 17 και τη 41. Ε, συγγνώμη, την 16, την 17 και τη 41. Φαντάζομαι ότι δεν πρόκειται για τη σωστή αιτιολόγηση. Το καταλάβατε αυτό, ότι πρόκειται για μια άλλη οδηγία. Κάποιο μπέρδεμα έγινε εκεί πέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σωστή η αιτιολόγηση που αναφέρεται εκεί. Πάντως λοιπόν για τη 16 τώρα, τη 17 και τη 41 μιλάει για 6 εβδομάδες υποχρεωτική άδεια μητρότητας. Ξέρω ότι ο ILO μιλάει για υποχρεωτική, αλλά εγώ νομίζω ότι εξαρτάται από τον καθένα, τι θέλει ο καθένας. Να μπορεί κανείς να επεκτείνει την άδειά του, αλλά να υποχρεώνουμε κάποιον κάποια γυναίκα έξι εβδομάδες αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού, κάποιος μπορεί να το θέλει, κάποιος μπορεί να θέλει περισσότερο, ε, κάποια άλλη γυναίκα μπορεί να μην είναι σε θέση να καθίσει τις έξι εβδομάδες. Γι' αυτό ελπίζω να υποστηρίξετε τη 16, τη 17 και τη 41 που θέλουν διαγραφή της υποχρεωτικής φύσης των ε, έξι εβδομάδων. Ευχαριστώ. Κυρία Σρέντερ και μετά η κυρία Στάουνερ. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να κοιτάξουμε αυτά τα οποία έθιξε και η συγγήτρια. Εκεί που αναφέρει ότι δεν καταλαβαίνει γιατί υπέβαλε τις τροπολογίες αυτές. Οι τροπολογίες αυτές ε, και η αλλαγή της οδηγίας για την προστασία της μητρότητας Αναφέρεται καταρχάς ε, στην ε, Οδηγία 2002-73 για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Αυτό αποτελεί την γενικότερη βάση και εξ όσων γνωρίζω το σημείο αυτό ακριβώς της υποστήριξης εκείνων που θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό ε, δεν τονίζεται επαρκώς στην οδηγία αυτή και ο λόγος είναι ότι θέλω να υπάρχει συμβατότητα και με την οδηγία κατά των διακρίσεων. Γιατί γνωρίζω κάποια παραδείγματα στην πράξη που ακριβώς αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν μπορούν οι μητέρες να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ αυτή την ε, ενίσχυση, αν θέλετε, για να υπάρχει συμβατότητα με την οδηγία κατά των διακρίσεων. Και αυτό ευθύς εξ αρχής. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό στην Ευρωπαϊκή και είναι σαφές μάλλον προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι σημαντικές αυτές ε, οι τροποποιήσεις γιατί καθίσατε σαφές ότι στην πραγματικότητα δεν είναι δυνατόν να περάσουν οι αλλαγές αυτές χωρίς να ασκηθεί πίεση. Ευχαριστώ κυρία Στάουνερ. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. να διορθώσω κάτι τυπικό. Με φρίκι μεν, αλλά να το πω στη γραμματεία ότι κατά λάθο λόγω του γραφείου του Τόμας Μαν αναφέρομαι κι εγώ ως ε, συντάκτρια της ε, όχι, όχι, όχι. Οι 38, 39, οι 44 και οι 47 είναι οι τροπολογίες αυτές ακριβώς που δεν συμφωνώ σε καμία περίπτωση με τον Τόμας Μαν. Ναι, μεν είναι από την ομάδα μου, αλλά είναι λάθος. Δεν είμαι συντάκτρια των γνωματοτήσεων, γιατί αυτό θα ήταν αντιφατικό με τις τροπολογίες που υπέβαλα. Γι' αυτό λοιπόν να παρακαλέσω τη γραμματεία την 38, 39, 44 και 47, από όσο είδα έτσι γρήγορα γρήγορα, να παρακαλέσω τη γραμματεία να διαγράψει το δικό μου το όνομα. Μία γενική παρατηρήση θα ήθελα να κάνω τώρα. Να παρακαλέσω την εισηγήτρια και περνώ στη δική μου τροπολογία υπαριθμών 15. Παρακαλώ λοιπόν την ε, εισηγήτρια να λάβει υπόψη ότι υπάρχουν κράτη-μέλη όπου υπάρχουν ε, και ρυθμίσεις γονικών αδειών ή αδειών ανατροφής, όπως αναφέρονται. Να το αναφέρει και αυτό. γιατί σκοπός της τροποποίησης της οδηγίας είναι οι μητέρες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αν και υποστηρίζω απόλυτα τους 18 μήνες, να μπορούν να επανέρχονται στο επάγγελμά τους. Αλλά υπάρχουν σίγουρα και χώρες όπου η νομοθεσία προβλέπει και η Γερμανία είναι μία από αυτές τις χώρες όπου η νομοθεσία προβλέπει άδεια για μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ανατροφή του παιδιού. Αυτό κάπως να αναφερθεί έστω στην οδηγία. Καταλαβαίνω φυσικά ότι υπάρχουν και άλλες ρυθμίσεις ε, οι οποίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να άπτονται τέτοιων ζητημάτων όπως οι γονικές άδειε, αλλά θα ήθελα να υποστηρίξετε την τροπολογία μου υπαριθμών 15. Νομίζω ότι θα ωφελούσε πάρα πολύ στο σύνολό της την οδηγία. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαντέρα, αφού ακούσαμε όλους τους ομιλητές, κυρία Μαντέρα για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πριν από οτιδήποτε άλλο, ευχαριστώ πολύ τους συναδέρφους για τις εξηγήσει. Όσον αφορά τις τροπολογίες 21 και 58, είχα κάποιες ανησυχίες Αναρωτιέμαι δηλαδή κατά πόσο εδώ είναι το σωστό μέρος στην οδηγία προκειμένου να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα. Γιατί έτσι κι αλλιώς πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχουμε προφυλάξει, έχουμε διατηρήσει. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Τώρα, στη συνάδελφο Λίν. Ειλικρινά δεν ε, μίλησα ακόμα για τις τροπολογίες της και γιατί. Διότι μετά τη συζήτηση είχα καταλάβει ότι έξι εβδομάδες είχα σαν στόχο να προστατεύσουν τη γυναίκα. Η γυναίκα έχει τη δυνατότητα. Το κράτος όμως πρέπει να εγγυάται, πρέπει να εξασφαλίζει την προστασία αυτή της γυναίκας. Να όλοι το δικαίωμα, όλες το δικαίωμα αυτό, αλλά αν θέλουμε να γυρίσουμε μέσα στη δουλειά μας, δικιά μας δουλειά. Ο νόμος πρέπει να εξασφαλίζει, να εγγυάται τη δυνατότητα αυτή. Αυτή η δυνατότητα πρέπει να διατηρηθεί ακόμη και αν η γυναίκα αποφασίσει κάτι διαφορετικό. Οπότε, ανεξάρτητα από την ατομική θέληση που έτσι κι αλλιώς προέχει, στόχος μας είναι η οδηγία να εγγυάται ότι διατηρείται η περίοδος αυτή των 6 εβδομάδων. Στην κυρία Στάουνερ τώρα. Η τροπολογία σας δεν μου δημιουργεί κανένα πρόβλημα η 15 διότι υπάρχουν πολλές προτάσεις, πολλές από αυτές πάνε προς την ίδια κατεύθυνση. Εξάλλου και εγώ στην πρώτη συζήτηση είχα πει ότι δεν μου άρεσε πολύ η οδηγία να συζητιέται χωριστά. Εγώ θα ήθελα σφαιρικά να συζητούσαμε το πρόβλημα, αλλά πάντως δεν έχω κανένα πρόβλημα με την τροπολογία σας αριθμός 15. Ευχαριστούμε. Έληξε η συζήτηση για αυτό το θέμα, συνεπώς θα ψηφίσουμε στις 31 Μαρτίου. Έληξε η συζήτηση λοιπόν για αυτό το θέμα προς το παρόν σήμερα. Περνάμε στην κοινή συζήτηση, σημεία 11 και 12, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία προαιρετικό πρωτόκολλο. Πάλι δηλαδή για τα άτομα με αναπηρίες. Εδώ Έχω συζητήσει με την κυρία Γέλεβα, την εισηγήτρια, και πρόκειται για συμβάσεις για τις οποίες τα κράτη-μέλη πρέπει να απαντήσουν με ναι ή όχι. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε τη θέση μας ή και να τη δώσουμε δεν μπορούμε να επηρεάσουμε ούτε τη σύμβαση ούτε το πρωτόκολλο. Συμφωνήσαμε λοιπόν για την εξής διαδικασία. Καταρχήν, σύνταξη ενός ψηφίσματος με μία δήλωση της Επιτροπής. Συνεπώς, ό,τι τροπολογίες υπάρχουν στη σύμβαση και στο πρωτόκολλο θα συμπεριληφθούν στο ψήφισμα. Και θα καθορίσουμε νέα προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών στο ε, ψήφισμα για τις 6 Μαρτίου. Αυτή λοιπόν είναι η πρότασή μου. Όταν θα εξετάσουμε το σημείο αυτό, όταν δηλαδή θα το ψηφίσουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι πρόκειται για την σύμβαση, για το πρωτόκολλο και για το ψήφισμα. Κυρία Γιάλεβα, έχετε το λόγο όμως, παρακαλώ. Благодаря, господин председателю. наи искам да благодаря на всички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 να πω κάτι στους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες και στις δύο εκθέσεις. Έχω λάβει 34 τροπολογίες για την ε, σύμβαση και 99 για το προαιρετικό πρωτόκολλο. Και όπως είπε ήδη και ο Πρόεδρος, πολλές από αυτές τις τροπολογίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν μη παραδεκτές λόγω της ε, διαδικασίας που έχουμε επιλέξει. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τη διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ήταν πάντα πολύ συνεπές στις προσπάθειές του να προωθήσει νομοθεσία υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες και να εξασφαλίσει τα δικαιώματά τους. Και όπως είπαμε και την περασμένη φορά, είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δίνει τη γνώμη του για μια σύμβαση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα συμφωνήσετε λοιπόν όλοι μαζί μου ότι θα πρέπει να πούμε κάτι παραπάνω από ένα απλό ναι, να δώσουμε δηλαδή απλώς το πράσινο φως στη σύμβαση. Αυτό είναι πολύ λίγο, δεν αρκεί. ήρθα σε επαφή με τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία σε πολλές χώρες και στη δική μου χώρα. Και από ό,τι φάνηκε, όντως περιμένουν να ακούσουν κάτι παραπάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ένα απλό ναι, από ένα απλό πράσινο φως. Είναι πολλές οι τροπολογίες, όπως είπα, και νομίζω ότι αξίζει να το συζητήσουμε το θέμα. Και γιατί υπάρχουν και πολλές τροπολογίες. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ακουστεί περισσότερο η φωνή μας για τη σύμβαση και για το πρωτόκολλο. Όταν η Επιτροπή μας άρχισε να δουλεύει πάνω σε αυτά τα δύο κείμενα, οι χώρες οι οποίες είχαν επικυρώσει την ε, σύμβαση και το πρωτόκολλο ήταν μόνο τέσσερις. Σλοβενία, Ουγγαρία, Ισπανία και Αυστρία. Τώρα, δύο επιπλέον χώρες έχουν ε, προσυπογράψει η Σουηδία και η Γερμανία. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, θα προτείνουμε ένα ψήφισμα. Θα έχετε λοιπόν στη διάθεσή σας το σχέδιο του ψηφίσματος και το ψήφισμα αυτό θα περιλαμβάνει ουσιαστικά όλες τις τροπολογίες που προτείνεται στην προφορική έκθεση και κάποιες ε, προτάσεις που κάνουν οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες. Καθώς και, κάθε, και κάποιες προτάσεις της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, των Γυναικών. Ελπίζω να ακούσω τα σχόλιά σας και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Σας ευχαριστώ βέβαια και για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ένας μου έχει δει το λόγο, ή μάλλον μία, και είναι η κυρία Λίν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για το έργο σας, κυρία Γέλεβα. Συμφωνούμε και εκφράζω την, ε, τις ευχαριστίες μου που ε, περιλάβατε και τις ε, τροπολογίες που είχα υποβάλει στο αρχικό σχέδιο χθες και τώρα θα μπουν στο ψήφισμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά ήθελα μόνο να πω. Σας ευχαριστώ. Ε, επιθυμεί κανείς άλλος να σχολιάσει. Εσείς κύριε Γέλεβα δεν θέλετε. Καλά λοιπόν. Τότε <clears throat> ολοκληρώνει τη συζήτηση. Α, ο κύριος Μα... Μπούσιλ Μάθιους. Δεν είμαι βέβαιος ότι υποθέτω σωστά, αλλά επειδή πρόκειται για ψήφισμα που με κάποιο τρόπο θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή, θα φέρει το όνομα της αρχικής συζήτησης, έτσι δεν είναι μαζί με άλλα ονόματα. Αλλά να είναι σαφές ότι ε, η κινητήρια δύναμη για το ψήφισμα είναι η κυρία Γέλεβα. αυτό ήθελα να επαληθεύσω την ιδέα μου αυτή. Σας ευχαριστώ. Διευκρινίστηκε λοιπόν αυτό το ερώτημα. Ψηφοφορία επί του θέματος θα γίνει στις 31 Μαρτίου και για το πρωτόκολλο και για το ψήφισμα. Προχωρούμε λοιπόν τότε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι η ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα. Κύριε Σίλβα Πενέντα, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Νομίζω ότι το αρχικό κείμενο ε, είχε εκπονηθεί τον Νοέμβριο πέρσι. Δεν γνωρίζαμε ακόμη τότε την έκταση της οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις της και στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Τους τελευταίους μήνες προστίθενται, συσσωρεύονται οι αρνητικές ειδήσει και αυτό επηρεάζει και τις 22 τροπολογίες τις οποίες έχω καταθέσει και άλλες μαζί με τον κύριο Σκομπάρ το κείμενο που θα υποβληθεί στους, υποβάλλεται τώρα μάλλον στους συναδέλφους, είναι πιο προσαρμοσμένο στις νέες τροποποιημένες ε, συνθήκες. Ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφους για τις περίπου 200 τροπολογίες που κατέθεσαν και τις οποίες εγώ ανέγνωσα προσεκτικά και μάλιστα μέσω των σκιωδών εισηγητών έχω υποβάλει και διάφορα κείμενα στις πολιτικές ομάδες ε, με την έννοια περισσότερο συμβιβαστικών τροπολογιών. Και γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι ε, είναι σημαντικό να εξεύρουμε κάποια ισορροπία, να θέσουμε σωστά κάποιες προτεραιότητες στον κοινωνικό τομέα. Βέβαια πρέπει να λάβω ε, οπωσδήποτε υπόψη ότι το βασικό είναι να ανακάμψει η ευρωπαϊκή οικονομία και σε αυτή την βασική ιδέα επανερχόμαστε και εν ώψη της ε, σοβούσης κρίσεως πρέπει να πούμε σαφώς ότι χρειαζόμαστε μια Ευρώπη όπου να ενισχυθεί η κοινωνική πολιτική. Αυτό είναι προφανές και από τα πιο σημαντικά θέματα. Διότι εν τέλει αυτό που μας απασχολεί είναι να διαφυλάξουμε την κοινωνική ειρήνη. Άρα δεν επιτρέπεται να μειώσουμε τις κοινωνικές δαπάνες. Πρέπει ε, μάλλον να αναδιαρθρώσουμε ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και να το κάνουμε πλέον αηφόρο. Την προηγούμενη εβδομάδα επέβαλα 18 προτάσεις συμβαστικών τροπολογιών στους διάφορους και οδησίτες. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν μάλλον θέματα στα οποία να μην μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμβασμό ώστε να διαμορφωθεί καλά το σχέδιο της εκθέσεως. Θα έρθω σε λίγες από αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες για παράδειγμα για την ιδεολογική σκέψη Γ, νομίζω ότι εκεί επιτυγχάνουμε ένα συμβιβασμό, ε, αφού πρόκειται για τα πιο ε, τροτά, τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, για τους πτωχούς. Είναι οι 19, ε, είναι οι 20 του κ. Λέιντε και άλλες τροπολογίες που αναφέρονται στα θέματα αυτά και εγώ έκανα μια προσπάθεια να τονίσω, εν πάση περιπτώσει δεν είμαι αντίθετος με την τροπολογία 41 της ε, κυρίας ε, Λίν, καθώς επίσης της κυρίας Κασιωτό, Κασιώτου και διαφορών άλλων τροπολογιών που κατευθύνονται λίγο πολύ στην ίδια κατεύθυνση. Επιθυμώ να επιτύχω να επιτύχω τα ίδια που ζητεί και στην 74 ο κ. Κρέμερς και ε, μπορούμε με την τροπολογία αυτή νομίζω να συνδυάσουμε και την 54 και 58. Επίσης την 75 και την 78. Όλα αυτά μπορούν νομίζω να, ε, όλα τα, τα, περιεχόμενα αυτά μπορούν να συγχωνευτούν σε ένα και νομίζω ότι έτσι θα είναι πλέον συνοπτικά. Με στόχο όπως είπα να επιτευχθεί μια ισορροπία. Έχω και την 91 του κ. Κρέμερς 82 Παπαδημούλη, ο Κούστασερ και ούτω καθεξής. Στην 9, συμβαστική 9, πρόκειται για την κοινωνική πολιτική και πώς αυτή μπορεί να συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή. Εκεί βάζω τις αεροπολογίες Κούστασερ και Σκομπάρ, την υπαριθμόν 75 δηλαδή. Στην παράγραφο 13 ε, αναφέρεται αυτή σε ενεργότερη συμμετοχή των εργαζομένων στην επιχείρηση. Υπάρχουν πάλι εκεί διάφορε τροπολογίε οι οποίε όλε μπορούν να συμπεριληφθούν σε μια ενιαία συμβιβαστική τροπολογία, όπω για παράδειγμα ορισμένε του κ. Μπούσιλ Μάθιου, η 117 λέει ντε. Ε, παράγραφο 14 αναφέρομαι στι ε, αρνητικέ επιπτώσει τη μεταναστεύσεω και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να συγχωνεύσουμε την 128, 130 και 137 δικές μου Ευχαριστώ και τον ε, κύριο Μπούσιλ Μάθιους για τις τροπολογίες που ίδιος έχει καταθέσει. Επίσης, ορισμένες άλλες τροπολογίες που επιθυμώ να συμπεριλάβω σε ένα νέο κείμενο όπως έχει διατυπωθεί και αυτό από τον κύριο Μπούσιλ Μάθιους. Ορισμένες άλλες τροπολογίες όπως η 183 και 153 της, ε, ε, ε, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών. Αναμένουμε και γνωμοδοτήσεις από άλλες επιτροπές, όπως την Επιτροπή Πολιτισμού. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους μου λοιπόν, ευχαριστώ και τους και και νομίζω ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με ιδιαίτερα θετικό τρόπο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κρέμερς και μετά ο κύριος Κουστάτσιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Το μήνυμα του συναδέλφου Πενέδα. Και εμείς, τουλάχιστον η ομάδα μας, σίγουρα συμφωνεί με τον στόχο του για να τα διατυπώσει όλα αυτά σαν ένα μήνυμα περί της κοινωνικής πολιτικής για να μην απειλείται αυτή. Συνεργαζόμαστε λοιπόν πολύ καλά. Οι κύριες προτάσεις που διατυπώσαμε αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη φιλοδοξία. Η Επιτροπή ήρθε το καλοκαίρι με την νέα κοινωνική ατζέντα, κάτι το οποίο εμεί βρήκαμε ότι έτσι κι ήταν πολύ αργά εκείνη τη στιγμή, ότι δεν ήταν αρκετό το περιεχόμενο έτσι καλώς έχουμε συζητήσει και άλλα πράγματα εδώ στην Επιτροπή μας, οπότε αυτά όλα δείχνουν ότι πρέπει να προσθεθούν και άλλα πράγματα στην κοινωνική αυτή ατζέντα. Για την αξιοπρεπή εργασία, για τα θέματα που έχουν να κάνουν με χαμηλές αμοιβέ, με τις λογικές συμβάσεις κλπ. κλπ. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε μπει στο σωστό δρόμο με τον συνάδελφο Πενέδα προκειμένου να υποβάλουμε τροπολογίες προς τη σωστή κατεύθυνση. Ένα πρόβλημα υπάρχει βέβαια με τη μετάφραση μιας τροπολογίας μου που μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις. Η 112 ζητάει από την Κομισιόν να ε, κάνει μια διάκριση από τη μια μεριά οι εργοδότες που αυτοποσχολούνται και από την άλλη μεριά εργοδότες που έχουν ε, ε, δικού τους εργαζόμενους. Η μετάφραση δεν έχει γίνει σωστά πάντα. Δεν όλες τις γλώσσες για αυτοαπασχολούμενους. Για μένα είναι ξεκάθαρο. Από τη μια μεριά έχουμε τους αυτοπασχολούμενους που είναι πραγματικά αυτοπασχολούμενοι που είναι ο άνθρωπος ορχήστρα κατά κάποιο τρόπο, ένας, και από την άλλη μεριά είναι ο επιχειρηματίας εκείνος που έχει εργαζόμενους στη γλώσσα μου, στα Ολλανδικά τουλάχιστον, δεν έχει μεταφραστεί όπως θα έπρεπε. Στα αγγλικά νομίζω ότι εγώ κατέθεσα αυτή την τροπολογία και δεν έχει μεταφραστεί καλά στα αγγλικά. Εν πάση περιπτώσει, ας το κοιτάξουν αυτό οι αρμόδιοι. Και να συζητήσουμε μετά για τις συμβαστικές ενδεχομένω τροπολογίες. Α, και μένα μου έχει συμβεί, να ξέρεις. Όταν είχα έκθεση για δικαστικές υποθέσεις λαβάς. Και τότε να ξέρεις ότι ορισμένες τροπολογίες δεν είχαν μεταφραστεί καλά στα σουηδικά. Ωραία. Τώρα, ο κύριος Κουστάτσα πρώτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με τις παρατηρήσεις του Ρολαλίσεντα, του κύριου Κρέμης, αλλά θα ήθελα να τοποθετηθώ αναφορικά με τις τροπολογίες του κυρίου Πινέδα που θεωρώ ότι αποτέλεσαν βελτίωση και νομίζω ότι στις συμβαστικές ε, προτάσεις σας έβαλε κάποια στοιχεία τα οποία με βρίσκουν σύμφωνο. Για κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τώρα θα ήθελα να τοποθετηθώ. Εκεί που αναφέρεται για την καταπολέμηση της ένδυας αναφορικά όλα τα άτομα τα οποία έχουν πληγθεί από την Ένδια. Λυπάμαι γιατί οι Ρωμά, οι μετανάστες, οι μετανάστες χωρίς χαρτιά δεν αναφέρονται. Ξέρουμε, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτοί είναι η πιο φτωχή. Αυτή είναι στον πάτο της κοινωνικής πυραμίδας. Και Πολύ απλά αυτοί κατηγορούνται τελικά και είναι η υποδοτουργία ή τράγοι για όλα όσα πάνε στραβά στην Ευρώπη. Είτε μιλώ για την Ιταλία, είτε μιλώ για την ε, Αυστρία. Αυτό είναι δραματικό. Αυτοί που δεν έχουν εκλογικό πρόγραμμα και τελικά καταδικάζουν και κατηγορούν τους ε, μετανάστες, αυτοί είναι τελικά που επιβραβεύονται στις εκλογές. Θα πρέπει λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φέρουμε ρητά ότι και για αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να υπάρξει πολιτική για την ενσωμάτωσή τους και σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της ένδυας. Για τη συμβαστική 2. Συμφωνώ. Στη Συμβιβαστική 1 θα προτείνω να κάνουμε και μία προφορική τροπολογία για την συμβαστική 2. Συμφωνώ. Ακόμα και αν δεν αναφερθούν τα προληπτικά μέτρα τα οποία εγώ αναφέρω ρητά, δεν είναι τόσο ουσιώδες. Στη συμβαστική 3 αντιμετωπίζω κάποιες δυσκολίες. Αυτό το θέμα της flexicurity, της ευέλικτης ασφάλειας, παρουσιάζεται ως πανάκια πολλές φορές αλλά πρόκειται για πανάκια από την πλευρά των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την ελευθερία, την κινητικότητα από πλευρά των επιχειρήσεων. Αλλά υπάρχει και η αντίθετη όψη του νομίσματος. Θα πρέπει η ίδια ευελιξία να υπάρχει και από την πλευρά των εργαζομένων και δεν υπάρχει. Εγώ θέλω να υπάρχουν βιώσιμες θέσεις εργασίας και αυτό θα ήταν πιο σημαντικό, θεωρώ, και δυστυχώς δεν συμπεριληφθήκε για τη συμβαστική 4, για την πρόταση αυτή. Έλεγα εγώ ότι δεδομένου του ελάχιστου μισθού αφαιρέσατε το ελάχιστος, ελάχιστος μισθός. Και αυτό έγινε σκόπιμα, γιατί όταν μιλάμε για την επιδότηση της ίδρυσης επιχειρήσεων, εντάξει. Είναι όμως υπερβολικά απλοϊκό να πούμε ότι αυτοί που αντιμετωπίζουν δυσκολίες φταίνε οι ίδιοι και να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Για τη συμβαστική 5. Συμφωνώ. Εγώ θα ήθελα να είναι πιο εκτενής βέβαια γιατί θα ήθελα να συμπεριληφθεί και η περιφερειακή και τοπική πτυχή, αλλά συμφωνώ και με αυτή την πιο συντεμημένη έκδοση της ε, τροπολογίας. Και το ίδιο μπορώ να πω και για την συμβαστική παριθμόν 6, για την ε, κοινωνική, βιώσιμη πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο. Συμφωνώ ε, με την πιο σύντομη αυτή διατύπωση του κυρίου Πινέδα. Συμφωνώ. Και σας ευχαριστώ κύριε Πινέδα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Λοίδου και μετά ο κύριος Μπούσιλ Μάθιου. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Σίλβα Πενέδα για τη δουλειά του. και για τις ε, απόπειρες συμβιβασμού νομίζω ότι θα φτάσουμε σε θέσεις πολύ γειτονικέ για να μην πω κοινέ. Είναι πολύ σημαντικό κάτι που είπε προηγουμένως, θα το τονίσω κι εγώ, το γεγονός ότι για πολλούς από εμά σε αυτή την Επιτροπή ένα από τα επόμενα βήματα της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να δημιουργηθεί μια πραγματική κοινωνική Ευρώπη όπου σε κάποιους τομείς πραγματικά δεν υπάρχει, απουσιάζει. Στην έκθεση λοιπόν που θέλουμε να υιοθετήσουμε Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Ο κ. Σίλβα Πενέρα είπε ότι δεν θα πρέπει να μειώσουμε τις ε, πιστώσεις, πολύ σωστά. Πολλά δε μάλλον που έχουμε μπει κανονικά σε αυτή την ε, τρομερή κρίση, θα πρέπει οι κυβερνήσει των κρατών μελών να καταλάβουν ότι ε, κάποιες πιστώσεις όπως αυτές για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση χρειάζονται αυτές οι πιστώσεις για να τα καταφέρουμε αυτά τα κονδύλια. Τώρα, περιμένω από κάποιους συναδέλφους με τους οποίους ήρθα σε επαφή κάποιες απαντήσεις για να δω αν θεωρούν ότι οι, δικές τους, οι δικές τους τροπολογίες έχουν ληφθεί υπόψη. Και όταν έχω τις απαντήσεις αυτές θα ενημερώσω αμέσως τον κύριο, αμέσως τον κύριο Σίλβα Πενέδα. Ένα τελευταίο σημείο που κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό, το ανέφερα δύο φορές τροπολογίες μου, το θέμα των κοινωνικών υπηρεσιών ε, καθολικής, ε, καθολικού ενδιαφέροντος. Καλό είναι να πούμε κάτι σε αυτό το κείμενο, ε, χωρίς να αναφερθούμε ειδικά σε αυτές, αλλά να κάνουμε μία έτσι, παραπομπή, αν θέλετε. Πρόεδρος, ο κ. Μπουσιμάθιος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή έχει όλα τα στατικά για να γίνει μια θαυμάσια και δυνατή έκθεση. Ευχαριστώ όλους όσους συνεισέφεραν με την εμπειρία τους και με τις απόψεις τους. Και πιστεύω ότι και οι απόψεις των υπολείπων πολιτικών ομάδων είναι πολύ σημαντικές. Συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο τα κοινωνικά θέματα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς φυσικά θα μας κατευθύνει ο εισηγητής. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους ότι για να είναι καλή αυτή η έκθεση, καλό είναι να μην είμαστε υπερβολικά άπλιστοι, να μην βάλουμε πολλά πράγματα μέσα εκεί, γιατί καλό θα ήταν να έχουμε μια μεγάλη διακομματική υποστήριξη για αυτή την έκθεση, παρά να έχει ο καθένας το δικό του κομματάκι ε, κάτι που θα δυσκολέψει την συνένεση. Καταρχάς, ε, η ελάχιστη μισθή, αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα γιατί έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Κάποια σχόλια για τους μισθούς πρέπει να γίνουν, για την, ε, για την ίση πληρωμή, για ίση εργασία κτλ. Αλλά είναι πολύ δύσκολο αυτό το θέμα και προσοχή πώς θα το προσεγγίσουμε. Κάτι άλλο. ε, οποιοδήποτε και αν είναι το θέμα, ξαφνικά ε, εμφανίζεται πάντα η οδηγία, γίνεται μια παραπομπή πάντα στην οδηγία για τους απεσπασμένους, α, απεσπασμένους εργαζόμενους. Δεν υπάρχει λόγος να τα, να τα δούμε αυτά τα πράγματα εδώ. Ε, Επίση, η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επίση, εμφανίζεται παντού. Έχει γίνει μαϊντανό. Ε, προσοχή, συνάδελφε. Α την κρατήσουμε απλή την έκθεση, απλή και πιο λακωνική, για να έχουμε όσο να τον πιο ευρεία α, συνένεση. Πρόεδρο. Θα θυμάστε την ε, συνένεση που είχαμε δημιουργήσει για την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Ε, Όντω έχετε δίκιο, υπήρχε συνένεση. Περίτω λοιπόν να αναφέρουμε ξανά αυτήν την οδηγία η κυρία Ταμασεύσκα. Η κυρία Κχαϊτή μετά και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν δύο πράγματα ουσίας και ένα τεχνικό που θέλω να θίξω παρακαλώ. Στις τροπολογίες επιστήνω την προσοχή μας στο θέμα των οικογενειών με πολλά παιδιά, στις πολύτεκνες οικογένειες, δεν ξέρω πώς είναι στις άλλες χώρες, αλλά εμείς στην Πολωνία το ψάχνουμε αυτό. Στην Πολωνία είναι μια ομάδα ανθρώπων, οι οικογένειες αυτές, οι πολύτεκνες, που χρειάζονται ειδικά μέτρα. Όταν έχουμε να κάνουμε με μόνο γονικές οικογένειες, πολύ συχνά είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι οι πολύτεκνες οικογένειες. Και γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι σφάλμα να παραβλέπουμε αυτή την κατηγορία οικογενειών, τις πολύτεκνες δηλαδή. Χρειάζονται βοήθεια για να μην βουλιάξουν στη φτώχεια. Γιατί τι εννοώ εντάξει δεν λέω ότι είναι τα περισσότερα παιδιά, αλλά εν πάση περιπτώσει πολλά παιδιά τελικά μεγαλώνουν κάτω από κακές συνθήκες, με ελάχιστη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, σε, με ελάχιστη πρόσβαση στις υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης κλπ. Το δεύτερο που θέλω να πω τώρα. Συμφωνώ με την πρόταση του κύριου Κωστάτζετ ότι είναι σφάλμα να χρησιμοποιήσουμε την ευελιξία και ασφάλεια σαν να πρόκειται για την πανάκια. Συμφωνώ μαζί του. Όμως, λυπάμαι που τελικά δεν πόρεσα να δω ούτε στα αγγλικά ούτε στα πολωνικά τις συμβαστικές. Τι να κάνουμε, εγώ στα γαλλικά δεν τα καταφέρνω και μόνο στα γαλλικά τις έχω. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Να είμαι σε μια επιτροπή και να μην μπορώ να διαβάσω τα έγγραφα, αυτό το βρίσκω ότι είναι απαράδεκτο. Πρέπει να υπάρχουν πάντα μεταφρασμένα τα έγγραφα στην αίθουσα, στις γλώσσες μας. Ευχαριστούμε. Κυρία Κρετή τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη από τους συναδέρφους επειδή έλειπα ήμουνα στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς για τις προφορίες εκεί. Συναντήθηκα και με την κυρία Κούνεβα την Επίτροπο που συμμετείχε στην Επιτροπή εκείνη. Γι' αυτό άργησε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεύτερον, θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον εισηγητή Σίλβα Πενέδα για το πνεύμα συνεργασίας και διαλόγου που επιδεικνύει. Έτσι καταφέραμε να μην έχουμε τελικά διαφορές μεταξύ μας. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφωνίες ορισμένα πράγματα, αλλά δεν είναι πολύ σημαντικά. Όπως έχουμε πει και νωρίτερα, στηρίζουμε κάθε συμβιβασμό που έχει σαν στόχο την απλοποίηση του κειμένου. Εμείς θέλουμε η έκθεση αυτή να είναι σαφής, να μην είναι πολύ μεγάλη και θέλω να ζητήσω και κάτι από την Επιτροπή μας. Υπάρχουν μερικές τροπολογίες που ο εισηγητή μα λέει να καταψηφίσουμε επειδή συμπεριλαμβάνονται ήδη στην γνωμοδότηση τη επιτροπή για τα Δικαιώματα της γυναίκα. Όμω μερικέ φορέ βλέπετε αγνοούμε πλήρω τι νομοδοτήσει της επιτροπή Δικαιωμάτων της γυναίκα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα ήθελα να μην απορριφθούν οι τροπολογίε αυτέ, να μην τι θεωρήσουμε ε, περιτέ και να μην απορρίψουμε τη θέση της επιτροπή Γυναικών. Υπάρχει μια σειρά τροπολογιών που έχει ως στόχο να απαλύνει κάπως την κριτική που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντάξει, εγώ είμαι αισιόδοξη και πιστεύω ότι θα βρούμε κάποια συμφωνία εδώ. Θα ήθελα όμως το πρόβλημα που έχει να κάνει με τους περισσότερους πολίτες να συμπεριληφθεί στην έκθεση. Ακόμα και αν τα κράτη αντιστέκονται όταν πρόκειται για τους ελάχιστους μισθούς, εμείς Έχουμε χρέο απέναντι στου πολίτε και ω Ευρωβουλευτέ πρέπει να το βάλουμε σαν προτεραιότητα το θέμα των μισθών. Ακόμα και αν δεν έχουμε αρμοδιότητε γι' αυτό και είναι τα κράτη. Εκπροσωπούμε εμεί του περισσότερου Ευρωπαίου πολίτε. Υπάρχουν και κάποιε βέβαια λεπτομέρειε. Ο Γιάνν Κρέμερ ήδη εξέφρασε την άποψη των σοσιαλιστών και εδώ είμαι αισιόδοξη και ελπίζω ότι θα βρούμε μια λύση. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ τον κύριο Σίλβα Πενέδα για την τόσο καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λίν. Ευχαριστώ κι εγώ. Είχαμε πολλές συζητήσεις μέχρι τώρα για την κοινωνική ατζέντα, για την ανεωνομένη ιδιαίτερα κοινωνική ατζέντα. Είχα κι εγώ έκθεση όπου είχαμε συμπεριλάβει πολλά από αυτά. Οι δύο αυτές ε, εκθέσεις έχουν κοινά σημεία. Συγχαρητήρια λοιπόν για τη δουλειά σας πάνω σε αυτή την έκθεση. Εγώ μπορώ να δεχτώ τους συμβιβασμούς που συμπεριλαμβάνουν και τις δικές μου τις τροπολογίες. Δεν ξέρω αν σας το είπα, αλλά ναι, τις δέχομαι αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες. Είναι εντάξει για μένα. Τώρα αυτό για τους ελέγχιστους μισθούς. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες εδώ που όντω μιλάνε, λένε ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν κάποια προγράμματα για τους ελάχιστους μισθούς και θα ρίνουμε τα κράτη-μέλη να έχουν μια πρόβλεψη για ελάχιστους μισθούς ή ελάχιστα εισοδήματα. Αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να συμπεριληφθούν οι περιπτώσεις των ανθρώπων που έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα. υπάρχει και νομοθεσία για, κατά των διακρίσεων που θα πρέπει να εφαρμόζεται. Αλλιώς, πώς να μιλάμε για ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα. Συνεπώς, γι' αυτό που λέμε να μην βάλουμε μέσα πράγματα τα οποία τελικά δεν θα στηριχθούν, ε όχι, αν αρχίσουμε και βγάζουμε πράγματα ουσιώδη για την ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα, η έκθεση αυτή θα καταλήξει πολύ χειρότερα από ότι αν τα αφήναμε μέσα. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Σίλβα Πενέιντα, λέει ο πρόεδρος, να πω κάτι για τον ελάχιστο μισθό που στις σκανδιναβικές χώρες εμείς όλα τα βάζουμε αυτά στις συλλογικές συμβάσεις και τους ελάχιστους μισθούς εντάσσονται στις συλλογικέ συμβάσεις. Αν λοιπόν περιλάβετε και τέτοια πράγματα, πρέπει να δείτε τι κάνουν και οι επιμέρους χώρες μέλη μέσα στις παραδόσεις τους. Εάν αυτά δηλαδή τα επιβάλλουν νομοθετικά ή εάν εντάσσονται στις συλλογικέ συμβάσεις των κοινωνικών εταίρων και ούτω καθεξής. Ο κ. Σίλβα Πενέδα πάντα πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τις συναδέλφους και τους συναδέλφους και για τα ευγενικά τους λόγια. Υπάρχουν ορισμένε τροπολογίε που δεν μπορώ να αποδεχτώ. Ορισμένε άλλε επιθυμώ να τις σχολιάσω. Βεβαίως όλες οι πολιτικές ομάδες έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες. Το ερώτημα είναι να περιλάβουμε όλες αυτές τις τροπολογίες και τους μετανάστες, τους νέους, τους γεροντότερους, τους άνεργους, τις γυναίκες, τις ε, παραμεθόριες περιοχές, τις ε, ε συμβάσεις εργασίας οι οποίες έχουν κάποιο στοιχείο αβεβαιότητας, την παιδική εργασία κτλ. Ε, ε, ο κατάλογος θα ήταν μακροσκελέστατος. Εκτιμώ τις ε, διάφορες αυτές ιδέες, αλλά εάν περιλάβουμε το σύνολο των στοιχείων αυτών θα καταστήσουμε την έκθεση εξαιρετικά δυσκίνητη ή, ή πάντως όλα αυτά θα μπορέσουν να μνημονευθούν άπαξ μόνο και δεν θα μπορέσουν να συζητηθούν ε, εν εκτάσει. Είναι σωστέ οι παρατηρήσει αυτέ, επαναλαμβάνω όμω, ότι αν τα περιλάβουμε όλα τα στοιχεία αυτά, ε, η έκθεση θα γίνει βαριά και δυσκίνητη. Θα πρέπει να δούμε ε, ποια από τι ομάδε αυτέ είναι ε, πλέον ευάλωτη από άλλε και ούτω καθεξή. Δεν νομίζω να προχωρήσουμε πολύ τότε. Άλλωστε τη συζήτηση αυτή την έχουμε κάνει στο παρελθόν κατά επανάληψη. Και είναι και θέματα αυτά τα οποία εντάσσονται σε άλλε εκθέσει. Είπαμε, η έκθεση να είναι σύντομη και αντικειμενική. Ας μην άρουμε πάλι αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Δεν ξέρω. Ίσως να μην είναι λάθος, αλλά ε, νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί τους σκόπους της έκθεσης όλες αυτές οι επαναλήψεις. Υπάρχουν θέματα δηλαδή τα οποία κατά επανάληψη έχουν συζητηθεί και κριθεί εδώ και προτιμώ να μην τα περιλάβω. Εκτός πια και αν κάποιο από τα παραλυπόμενα τα δικά μου κριθεί στη συζήτηση τόσο σημαντικό ώστε να πρέπει να το περιλάβω. Και υπάρχουν και κάποιες διατυπώσεις οι οποίες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλες εκθέσεις και τις επαναφέρουν εδώ οι συνάδελφοι. Εμείς θέλουμε να, όμως να καινοτομήσουμε κιόλας λίγο εδώ. Ωστόσο, ε, σε ορισμένα θέματα θα επανέλθω σε κάποιες ε, λύσεις οι οποίες έχουν αποδείξει την αξία τους, όπου κάθε χώρα μέλος έχει επιλέξει τις λύσεις της, δεν μπορούμε εμείς να υπαγορεύσουμε άνωθεν. Θα γράψουμε λοιπόν τότε ότι ε, σύμφωνα με τις συνηθισμένες διαδικασίες που ισχύουν στην τάδε χώρα. για τον κύριο Λεϊντε, για την κοινωνική πρόνοια. Ε, και εδώ έχει υπάρξει ε, σχετική έκθεση και έχει προτείνει ειδικά μέτρα. Αλλά κάπου ε, θα έπρεπε να μνημονευτεί μέσα στην έκθεση. Για τα άλλα θέματα τώρα. Χωρίς να θέλω να τοποθετηθώ επί όλων των σημείων. Νομίζω πάντως ότι με διμερείς συζητήσεις μπορώ να ε, μπω σε λεπτομέρειες και να συζητήσω με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Με αυτή την ε, γνωμοδότηση, την οποία θα ψηφίσουμε στις 31 Μαρτίου, δηλαδή στην επόμενη συνεδρίαση, κλείσαμε και το σημείο, τη συζήτηση το σημείο 13. Και πάμε στο τελευταίο σημείο της σημερινής ημερήσιας διάταξης που αφορά την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας. Η κυρία Λάμπερτ είναι η συγγήτρια. Ευχαριστώ. Μερικές φορές έχουμε την αίσθηση ότι ξαναβλέπουμε το ίδιο έργο, ξανακάνουμε τις ίδιες συζητήσεις που είχαμε κάνει. Το πλαίσιο, θα το θυμάστε, είναι το να απαντήσουμε στην ε, σύσταση της Κομισιόν. Το Συμβούλιο έχει επίσης συζητήσει τη σύσταση αυτή και αφορά το θέμα αυτό την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας. Πρέπει να εξετάσουμε διάφορους τομείς που η Κομισιόν και το Συμβούλιο έχουν επιλέξει. Είχαμε αρχικά πάνω από 100 τροπολογίες, οι οποίες ε, εμπλουτίζουν, ε, μακραίνουν την ε, έκθεση. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους. Υπάρχουν πάντως ένα ή δύο θέματα που είναι αμφιλεγόμενα, δεν θα σε εκπλήσει αυτό. Ορισμένα από τα θέματα αυτά ε, συζητήθηκαν και για την έκθεση Σίλβα Πενέδα. Το ένα από αυτά, τα θέματα, αφορά το ελάχιστο εισόδημα, την υποστήριξη του ελάχιστου εισοδήματος, τον ελάχιστο μισθό και σε αυτή την έκθεση είναι εκ των όν αυτό το θέμα γιατί είναι βασικό συστατικό της ε, σύστασης της Κομισιόν το ελάχιστο εισόδημα. Επομένως κάπως θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτά που πρότεινε η Κομισιόν. Ε, το πιο αφιλεγόμενο θέμα είναι η παράγραφος 6, όπου γίνεται λόγος για, την, για μια οδηγία για αυτό το θέμα. Θα πρέπει να βρούμε κάποιο συμβιβασμό γύρω από αυτό το θέμα. Υπάρχουν μια σειρά από εναλλακτικέ. Ανάλογα με το τι εστίαση θέλουμε να έχουμε. Ε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το Ευρωπαϊκό Έτος Εξάλληψης της Στόχιας 2010. Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Ε, ίσως αυτές θα πρέπει να ψάξουμε παρά να βρούμε συμβιβασμό συγκεκριμένο. Τώρα κάτι άλλο. Για θέματα Έχουμε από τη μία το ελάχιστο εισόδημα. Υπάρχουν άλλα θέματα, τα θέματα ερεσιμότητας. Δηλαδή, τι επιδόματα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να... Συγγνώμη, δεν διαβάζω τις, σωστά τις α, σημειώσεις μου. Ορισμένοι πιστεύουν ότι η αιρεσιμότητα είναι σημαντική και ορισμένοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να την προσεγγίσουμε με προσεκτικό, με προσεκτικό τρόπο, ειδικά όταν ε, βρισκόμαστε σε περίοδο ισχνών αγελάδων. Είναι πολύ πιο δύσκολο κάποιο να βρει τότε δουλειά. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε συμβασμό γύρω από την ε, παράγραφο 5, δηλαδή τι εντάσει ανάμεσα στα, στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και τι ευκαιρίες απασχολησιμότητας υπάρχουν το θέμα της πρόσβασης στις ε, υπηρεσίες ποιότητας στην παράγραφο 13 και στο θέμα της ε, κατάργησης των διακρίσεων στην παράγραφο 15. Νομίζω ότι και εκεί θα μπορούσε να υπάρξει ένας ε, συμβιβασμός που να συγκεντρώσει την πλειοψηφία. Επίσης την παράγραφο 22 για τον οδικό χάρτη και το πώς θα προχωρήσουμε. Οι περισσότερες από τις τροπολογίες μπορούν να γίνουν αποδεκτέ από μένα χωρί κανένα πρόβλημα. Ίσως όμω θα πρέπει να βρούμε είτε συμβιβασμού ούτω ώστε να έχουμε μία παράγραφο ή αλλιώς μία παράγραφος να είναι η βασική παράγραφος Και εφόσον σας ικανοποιεί αυτή η βασική παράγραφος, ε, όσοι έχετε σχετικές τροπολογίες, να αποσύρετε τι τροπολογίε αυτέ για να μην προσθέσουμε και άλλε παραγράφου. Ε, τώρα κάτι που έλεγε και ο κύριο Σίλβα Πενέδα για το θέμα των ε, ευπαθών ομάδων ε, και το κατά πόσο θέλουμε να τι ονομάσουμε αυτές τις ε, ομάδε ή αν θα θεωρήσουμε ότι συμφωνούμε για ποιε είναι αυτέ οι ευπαθεί ομάδε γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει και το αφήνουμε έτσι. τι αναφέρουμε απλώ γενικά. Είναι θέμα δικό σα τη επιτροπή, ό,τι θέλετε. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε είναι τι γίνεται με την χρήση του Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Περιφερειοποίησης, ε, Παγκοσμιοποίησης, συγγνώμη, ε, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη. Ε, έχουμε τέτοιες εκθέσεις, έχουμε την κοινωνική ατζέντα, ίσως καλύτερα εκεί να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. παρά στο σημείο που μας απασχολεί εδώ. Υπάρχουν και διάφορα άλλα θέματα τα οποία επανέρχονται, τα οποία υπήρχαν σε άλλες εκθέσεις. Εδώ υπάρχει μια δυσκολία για μένα ως εισηγήτρια. Γιατί υπάρχουν πράγματα που πραγματικά τα υποστήριξα και τα υποστήριξα και τα πρώτο συζητήσαμε. Παραδείγματος χάρη να καταγράψουμε την κοινωνική πραγματικότητα κτλ. Αλλά να σας ρωτήσω, Επιτροπή, να δούμε ποιες είναι ε, οι τροπολογίες που αφορούν την κοινωνική ένταξη, παρά να γενικολογούμε και να κάνουμε αναφορές σε διάφορα πράγματα, ε, όπως παραδείγματος χάρη ποιότητα της ε, πολιτικής ασύλου. Περί αυτού πρόκειται λοιπόν. Γενικώ πώ μπορώ να δεχτώ τι περισσότερε ε, τροπολογίε, αλλά θα πρέπει να κάνουμε κάποιε επιλογέ σε ό,τι αφορά την ορολογία, ακόμη και την ε, φιλοσοφία τη έκθεσή μα. Δηλαδή, αν πιστεύουμε ότι ένα ελάχιστο εισόδημα που μα επιτρέπει να ζούμε αξιοπρεπώ είναι το βασικό θέμα, ή αν θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια υποστήριξη του εισοδήματος. Ε, και πώς θα υποστηρίξουμε το εισόδημα αν κανείς έχει μόνο αυτό ας πούμε. Ίσως είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με τις διακρίσεις. Αυτό και το θέμα της αιρεσιμότητας. Αυτά και σε ευχαριστώ συνάδελφοι για τις τροπολογίες ε, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αποδεκτές. Σα ευχαριστώ. Έχουμε στον κατάλογο των ομιλητών την κυρία Μιλίν. Καταρχά ευχαριστώ. σα ευχαριστώ και για το έργο σα Και την παράγραφο 6 έχετε δίκιο. Θα αποτελέσει πρόβλημα. Εγώ υπέβαλα τροπολογία για την παράγραφο 6 και για το ελάχιστο εισόδημα μπορεί να συγκεντρώσουμε την επιστόριξη των συναδέλφων, γιατί δεν μιλάμε για ένα ελάχιστο εισόδημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μιλάμε για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών αναφορικά με τα θέματα ελάχιστου εισοδήματο και ίσως έτσι να μπορέσουμε να συνενώσουμε διάφορες πλευρές της συζήτηση πίσω από την πρόταση αυτή. Η 54 ήταν η τροπολογία μου αυτή, αν θυμάμαι καλά, που ανέφερε Α, όχι, δεν ήταν η 54. 54. Θα τη βρω, θα τη βρω τέλο πάντων. Και επίσης ε, υπέβαλα πολλές τροπολογίες για τους ανάπηρους και τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το ενόπνευμα, γιατί αυτό αποκλείει φυσικά τα άτομα αυτά από την αγορά εργασίας. Κάτι άλλο που τονίζω με τις τροπολογίες μας για την ηλικία υποχρεωτική συνταξιοδότησης. Πολύ σημαντικό και αυτό και θα πρέπει να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη αναφορικά με την ηλικία συνταξιοδότησης, αλλά η υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης νομίζω ότι αποτελεί λανθασμένο μέτρο. Για αυτά που αναφέρετε για τα άτομα που φροντίζουν άλλα άτομα. Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε μία παράγραφο και για αυτούς. Να συνενώσουμε πολλές από τις τροπολογίες που υποβλήθησαν για τα άτομα αυτά. Καλή ιδέα. Για τους ετούντες άσυλο και για τη δυνατότητά τους να εργαστούν. Νομίζω ότι και πάλι θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Δεν μπορούμε να υπαγορεύσουμε οτιδήποτε στα κρατημέλη, αλλά προφανώς είναι σημαντικό οι ετούντες άσυλο να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν. Γιατί σε πολλές χώρες αποκλείονται από την αγορά εργασίας και καλό θα ήταν να υπάρχει κάποια αναφορά. Ναι, συγγνώμη αν θέλετε. Γιατί γίνεται και μία συζήτηση εξ αριστερών μου. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τους ετούντες άσυλο και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ξέρετε τι τροπολογίες έχω υποβάλει και στο παρελθόν έχουμε συνεργαστεί άψογα Είμαι λοιπόν αισιόδοξη ότι θα καταφέρουμε να βρούμε συμβαστικές προτάσεις και για τις τροπολογίες αυτές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο μικρές παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Καταρχάς, εμείς ως σοσιαλιστές ασφαλώς και θα υποστηρίξουμε τις προτάσεις αναφορικά με το ελάχιστο εισόδημα το σύστημα που θα ακολουθηθεί είναι κάτι το διαφορετικό, αλλά εμείς σίγουρα θέλουμε να συμπεριλάβουμε αυτή την ιδέα. Δεύτερο στοιχείο. Υπάρχει ένας ε, τομέας στον οποίο θίγουν πολλοί συνάδελφοι στις τροπολογίες τους αναφορικά με την είσοδο στην ε, αγορά εργασίας και υπάρχει και ένα πολύ συγκεκριμένο στοιχείο, το στοιχείο της επαγγελματικής κατάρτισης, της διαβίους μάθησης κτλ. Αυτό θεωρώ ότι θα έπρεπε να τονιστεί λίγο παραπάνω. Υπευλήθησαν σχετικές τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση και ασφαλώς και θα τις υποστηρίξουμε και εμείς αυτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λάμπερτ. Λάμπερτ. Παίρνει το λόγο λοιπόν για να κάνει τη σύνοψη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και την Λίσλιν για τις τροπολογίες που υπέβαλε. Ναι, και σίγουρα θα καταφέρουμε να βρούμε συμβιβαστικέ λύσεις. Και χάρηκα που άκουσα την ε, στάση των σοσιαλιστών για αυτά τα βασικά θέματα. Έχετε δίκιο, πρόκειται για θέματα τα οποία μπορούμε να τα ενισχύσουμε. Και κάτι άλλο που ήθελα να τονίσω εξ αρχής. Έχουμε αρκετές τροπολογίες πλέον για τον ρόλο των τοπικών αρχών. Γιατί πρόκειται για ένα στοιχείο το οποίο ναι. τονίστηκε σε δύο-τρεις τροπολογίες. Το είχαμε υποτιμήσει το στοιχείο αυτό και θα θέλαμε όντως να το υπογραμμίσουμε πιο έντονα. Άρα ναι, θα δεχτώ αυτές τις τροπολογίες για το θέμα αυτό και θα υποβάλω και εγώ κάποιες σχετικές ίσως και να ευχαριστήσω και την κυρία Παναγιωτοπούλου που υποστήριξε κάποιες από τις τροπολογίες αυτές οι οποίες ε, το έκανε μάλλον και με πολύ, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα γιατί ίσως κάποιοι συνάδελφοι να χρειάστηκαν πιο πολύ χρόνο από τα 30 δευτερόλεπτα που είχαμε στη διάθεσή μας. Αλλά είμαι σίγουρη ότι τελικά θα καταλήξουμε σε μια λύση την, η οποία θα υποστηριχθεί από όλου. Ευχαριστώ. Τελειώνει η συζήτηση για αυτό το σημείο της ημέσιας διάταξης. Θα ψηφίσουμε στις 31 Μαρτίου και για αυτό το σημείο. Και τώρα, πριν τελειώσουμε, είχαμε σκεφτεί ότι θα πρέπει σήμερα να κάνουμε μια συνεδρίαση των συντονιστών. Μια και διεκπαιρέσαμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τόσο γρήγορα, χρησιμοποίησαμε την γραπτή διαδικασία. Ε, Επομένως δεν θα γίνει συνεδρίαση των συντονιστών. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σημείο στη μέση διάταξη, εφόσον δεν θα κάνουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. Α, ο κ. Μπούσιλ Μάθιος. Να δείξουμε ότι ενδιαφερόμαστε για τα προβλήματα της Προεδρίας. Πριν από λίγο ε, η, η, η Κομισιόν ε, ακύρωσε την ε, ρήτρα για το... για το φως του ήλιου. Ε, μήπως θα πρέπει να τη φέρουμε ξανά σε ισχύ αυτή την ε, ρήτρα ε, για την προστασία των δικών σας ματιών, έτσι, για να σας, να σας δείξω πόσο ενδιαφερόμαστε για τα μάτια της Προεδρίας. Μπορούμε να Φωτίζουμε όλους σας, όχι μόνο εμάς, όλους σας, για να μην υποφέρει κανένας. Αν είχαμε την κατάλληλη τεχνική θα μπορούσαμε να, φωτίσουμε, να φωτίζουμε ένα ή δύο άτομα τη φορά, ε, αυτούς που μιλάνε δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να το κάνουμε τελικά από ό,τι μου είπαν. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ κύριε Μπουσκημάθης που ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για την Προεδρία. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 30 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και Τρίτη 31 Μαρτίου. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή βοήθεια. Τελειώνει η συνεδρίαση εδώ.